good morning. We continue the meeting of the subcommittee and um, I must say that we had a very... Καλημέρα, λέει Πρόεδρος. Πάλι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση χθε που μιλήσαμε για τα νέα μέσα, τεχνολογία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχαμε όλου αυτού του εξαιρετικού ειδικού, άλλου εμπλεκόμενου, την Nokia, Siemens, Siemens, από την Google και και Επομένω ήταν πάρα πολύ καλή η ακρόαση και επίση παρουσίασε πάρα πολύ ενδιαφέρον η ακρόαση για το πώ έχει η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στον αραβικό κόσμο με το Freedom House. Αλλά βέβαια ήταν και πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσα και η εκδήλωση μετά που ακολούθησε με του ακτιβιστέ από, από Συρία, Αίγυπτο και επίση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η ομιλία του γιου του Αλ Μαλαχός που είναι ακτιβιστής που είναι φυλακισμένο στην Δαμασκό. Και επίσης θα πρέπει να κάνουμε και άλλες προσπάθειες μήπως απελευθερωθεί. Για να δούμε τώρα τι προβλέπει το πρόγραμμα γιατί έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές. Έχουμε την ώρα των ερωτήσεων προς την Κομισιόν. Η πρώτη ερώτηση είναι από την κυρία Αντρικένε την Αντιπρόεδρο και αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μεξικό. Θέλετε, όχι δεν θέλετε. Ωραία. Τότε ευθύ αμέσω ο λόγο στην Κομισιόν για τι απαντήσει. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα σας μιλήσω για το Μεξικό, γιατί στην αρμόδια ενική διεύθυνση έχω εγώ αυτό το τμήμα. Τζανφράνκο Μπουκίκη ονομάζομαι και εγώ έχω το, την υπηρεσία, το, το γραφείο που ασχολείται με το Μεξικό στην Ρελέξ. Ευχαριστούμε την αξιότιμη κυρία Βουλευτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μεξικό. είμαστε ενήμεροι για αυτή την κατάσταση όπως μας τα είπε η κυρία βουλευτή, και παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα με προσοχή και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό. στι συναντήσεις πολιτικού διαλόγου με το Μέξικο. αυτά τα συζητούμε τακτικά και το είπαμε και στη συνάντηση κορυφή την πρόσφατη. Και το Μεξικό έχει χαιρετήσει το ότι έχουμε τέτοιο διάλογο δίμερη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρώτη δε συνάντηση σχετικά έγινε στις 12 Πέμπτου 2010 ή στο Μεξικό όπω αναφέρθηκε. Και σε αυτή την συνάντηση καλύψαμε πάρα πολύ σημαντικά θέματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίω τη χρήση στρατιωτικών και, αστυνομικών όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, τους ακτιβιστές και ήταν νομίζω ευκαιρία να τα πούμε με ειλικρίνεια όσον αφορά ε, κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα για το Μέξικο. Επίσης έτσι μπορούσαμε να προτάξουμε τις θέσεις της Ένωσης και τονίσαμε το ότι θα πρέπει πλήρως να διερευνηθούν οι καταπατήσεις των δικαιωμάτων από τα σώματα ασφαλεία και το στρατό. Επίση είπαμε ότι προβληματιζόμαστε γιατί σε αυτέ τι περιπτώσει έχει πληφθεί μόνο και αποκλειστικά η στρατιωτική δικαιοσύνη. Απειλέ, ανθρωποκτονίε, βάρο ακτιβιστών και έχουμε και τι περσινέ δηλώσει τη ΕΕ για του ε, ε, για τους δημοσιογράφους που φωνεύτηκαν φέτος αλλά και κάποιους άλλους που είχαν υπεραμυθεί του κεραίου και είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει σε ένα διπλωματικέ αρχέ, ώστε να εφαρμοστούν κατευθυντήριε γραμμέ για να αυτοκινητά στο Μεξικό. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με του ακτιβιστέ στην Τιχουάνα, του δύο ακτιβιστέ. Επίση θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα προστασία. Το Μεξικό τώρα, πλευρά του τι είπε, ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί μια ομάδα εργασία ώστε να δούμε σε συγκεκριμένε περιπτώσει, συγκεκριμένα μέτρα σε σχέση με αυτού του ακτιβιστέ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε παρά να συμφωνήσει όσον αφορά δε τις ε, απειλές και ανθρωποκτονίες της βάρος των δημοσιογράφων. Ε, ο Μεξικό συμφώνησε ότι θα προβεί σε κάποιες κινήσεις και παραδέχτηκε ότι χρειάζεται να γίνουν βελτιώσεις. Για το πιστότερο στην Οαχάκα οι έχουν επιληθεί και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να προσάγουν ενώπιον της δικαιοσύνη του ε, ενόχους. Μόλις αυτή τη βδομάδα είχαμε τους εκπροσώπου της αντιπροσωπεία σε σχέση με την ΟΑΧ. Και ε, η, η Ρελέξ ήρθε σε επαφή με τον κύριο Σπάτσα και σε σχέση με το, τον φόνο της ε, κυρίας Καρίνια επαναλάβαμε εμείς το ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις σχέσεις με τρίτες χώρες. Οι σχέσεις Ένωση και Μεξικού αποσκοπούν στο να προαχθούν οι κοινέ αξίες, αλλά δεν είναι αποκλειστικά αυτός ο στόχος μας. Πρόκειται για στρατηγικό εταίρο. Και όλα τα θέματα θα πρέπει να θίγονται και στα πλαίσια Αυτά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε ένα κοινό εκτελεστικό πρόγραμμα το οποίο στις 16 Πέμπτου στη συνάντηση κορυφής εγκρίθηκε στις νοικομίγες και η ΜΕΝ και η ΔΕ είπαμε ότι έτσι έχουμε τρόπο θεμένη αξία σε αυτήν την τόσο σφαιρική και ολοκληρωμένη σχέση. Οπότε έτσι θα προωθήσουμε τα κοινά συμφέροντα, ενδιαφέροντα, αξίες, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία. Προσπαθεί λοιπόν να υποπλέψει να παρακολουθήσει εξελίξει με ό,τι μέσα έχει διαθεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό με χαρά τη συμμετέχει σε τέτοιε επαφέ και συναντήσει και θέλουμε να έχουμε τακτέ επαφέ με ε, τις κοινέ κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Κυρία Χαντρικέν, έχετε κάποιε παρατηρήσει ή ερωτήσει. Ναι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σα τα πω όμω λιθουανικά σήμερα. Э, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει κάποιες πληροφορίες, οι οποίες όμως θα πρέπει να συμπληρωθούν από συγκεκριμένες, πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Ποια είναι η στάση της μεξικανικής κυβέρνησης, ποια είναι τα μέτρα τα οποία έχει πάρει ήδη η μεξικανική κυβέρνηση εναντίον των δολοφονιών εις βάρος των δημοσιογράφων. Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση της πόλης του Μεξικού η κατάσταση έχει ξεφύγει. Οι πληροφορίες ε, που έχουμε σχετικά με την πίεση που ασκείται στους δημοσιογράφους δείχνουν μια παράδεκτη κατάσταση, ιδιαίτερα σε μια χώρα η οποία θέλει να είναι στρατηγικός εταίρος και οι στρατηγικοί εταίροι μας πρέπει να μοιράζονται μαζί μας τις κοινέ αξίες. Θα ήμουν ευγνώμων λοιπόν αν ο εκπρόσωπος της ε, Ευρωπαϊκής μπορεί να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Ένα μόνο πράγμα να συμπληρώσω. Είμαι αναπληρώτρια στην αντιπροσωπεία για το Μεξικό και θα ήθελα να προκαλέσω μια ακρόαση στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό και των δολοφονιών των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων και την κατάσταση επίσης στις φυλακές του Μεξικού η οποία είναι φρικτή, δεν μπορούμε να σιωπούμε πλέον. Ευχαριστώ κύριε Αντρικίενα. Ο εκπρόσωπος υπηρεσίας της Κομισιόν για το Μεξικό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως σας είπα προηγουμένως, Είχαμε μία ειλικρινή θα έλεγα συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα και για άλλα θέματα κατά τη διάρκεια του πρώτου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Μεξικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ξεκάθαρη εκφράζοντας συγκεκριμένες ανησυχίες γύρω από τα θέματα που θίξατε και η μεξικανική πλευρά έδειξε ιδιαίτερα πρόθυμη, κατανοώντας και ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες μας. Εξηγήσαμε τις ανησυχίες αυτές και την παρουσία του Υφυπουργού Γκόμες Ρομπρέδο πρότεινε την δημιουργία μιας ομάδας εργασίας. Μια ομάδα εργασίας η οποία θα ερευνήσει το θέμα στα πλαίσια της οποίας θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών είπαν ότι επιθυμούν να ξεκινήσουν επαφές μαζί μας για συγκεκριμένες περιπτώσεις, για συγκεκριμένες ενέργειες και αναφέρθηκε μάλιστα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών σε περιπτώσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη ειδικότερα για τους δημοσιογράφους. Έγινε μία παρουσίαση από τον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα για τις ενέργειες εις βάρος των δημοσιογράφων. Υπάρχει δηλαδή μια συγκεκριμένη υπηρεσία που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Και θα μας ενημερώνει για τις ε, Εξελίξει στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα για την δολοφονία τον μήνα Ιανουάριο τριών ε, δημοσιογράφων. Δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης όμως. Υπήρξε παρόλα αυτά μια αίσθηση ότι η κυβέρνηση παίρνει μέτρα για να ερευνήσει σε βάθος αυτές τις ε, πράξει ει βάρος των δημοσιογράφων. Δεν υπήρξε αναφορά όμω σε συγκεκριμένα μέτρα, σε συγκεκριμένε δράσει. από πλευράς των Μεξικανών. Ολέ. Απλά μας έδωσαν την αίσθηση ότι λαμβάνουν υπόψη σοβαρά τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έθεσε το θέμα της δολοφονίας της Μπέτη Καρίνιο και της Διάκοβα στα πλαίσια αυτού του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχω στείλει ε, επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομίζω ότι είναι μια υποδειγματική περίπτωση η δολοφονία αυτών των δύο γυναικών δημοσιογράφων που δείχνει την ατιμορρησία η οποία σοβεί αυτή τη στιγμή στην Οαχάκα. Ξέρουμε ότι ο υπόκοσμος συνεργάζεται με κάποιες τοπικές ελίτ και έτσι δεν προχωρούν οι διώξεις και οι δίκες και ε, γενικά οι κυρώσεις εις βάρος των παρανόμων. Υπάρχει ανάγκη να προστατευθούν επίσης και ε, η ανθρωπιστική βοήθεια που θα αποσταλεί ε, στους ηθαγενείς στην περιοχή του Σαν Χουάν Κοπάλα της Οαχάκα. Ξέρετε ότι ο Όμαρες Πέρσα, τον οποίο συναντήσαμε χτες, ήταν μαζί μας εδώ και συζητήσαμε το θέμα μαζί του και πολλοί πιστεύουν από αυτήν την ε, κοινότητα των Ινδιάνων ότι απειλούνται σωματικά. Και γι' αυτό θα πρέπει να, να πιέσετε τις αρχές του Μεξικό City έτσι ώστε να προστατεύσουν τα δικαιώματα και την ίδια την επιβίωση αυτών των Ινδιάνων. Μάλιστα Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Το έχουμε ήδη συζητήσει με τις Μεξικανικές Αρχές έχουν ζητήσει από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ε, ευρωπαϊκές ε, υπηρεσίες ε, ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα πρέπει να υπάρξουν ειδικέ θεωρήσεις και άδειε για να πάνε στην περιοχή. Ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση, η διασφάλιση ακριβώς των όρων ασφαλούς διέλευσης είναι ευθύνη ε, των μεξικονικών αρχών και οι αρχές, ε, η υπηρεσία μάλλον, η αντιπροσωπεία μας στην πόλη του Μεξικού παρακολουθεί τις ενέργειες των μεξικανικών αρχών. Αύριο προβλέπεται μια συνάντηση ανάμεσα στον υπεύθυνο της αντιπροσωπείας μας εκεί με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Είχαμε μια συνάντηση την Τρίτη με τους δικηγόρους των θυμάτων έχει τεθεί το πρόβλημα στις ομοσπονδιακές αρχές στον προηγούμενο διάλογο που είχαμε. Οι πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενημερώσουν ε, τους ε, πολίτες τους που συμμετέχουν στην αποστολή αυτή για τους κινδύνους, το υψηλό επίπεδο ε, κινδύνου και θα τους ενημερώσουν για τις ειδικές βίζες που θα πρέπει να ζητηθούν από τις Μεξικανικές Αρχές. Αυτά είναι τα προβλήματα έτσι όπως τα αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μπορούμε να περάσουμε στη δεύτερη ερώτηση. Η κυρία Κιλ Νίλσεν. Για τα δικαιώματα των ηθαγενών της Δυτικής Παπούας Θέλετε να επαναλάβετε την ερώτησή σας ή να ζητήσουμε από την Επιτροπή να απαντήσει. Το ερώτημα είναι σαφές. Αναφέρομαι ε, στους κατοίκους της Δυτικής Παπούα. Το θέμα όμως αφορά γενικότερα τα δικαιώματα των ηθαγενών. Και μετά την απάντηση της Επιτροπής ε, θα δω αν θα πρέπει να επανέλθω. Η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Κιλ Νίλσον σχετικά με τη σημαντική της ερώτηση για τα δικαιώματα των ηθαγενών. Ο συνάδελφος Πέδρο Μαρτίνες Βάργας θα σας μιλήσει για τη συγκεκριμένη περίπτωση της Ινδονησίας και της Δυτικής Παπούα. Σχετικά με τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να σας περιγράψω ποια είναι η πολιτική την οποία ακολουθούμε. Τα θέματα των ηθαγενών πληθυσμών είναι αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής μας πολιτικής, όπως και η δήλωση των Ηνωμένων Εθνών του 2007 για τα δικαιώματα των ηθαγενών λαών είναι το βασικό, η βασική μας αναφορά. Όπως λέμε σε περίεργα αγγλικά, προσπαθούμε εμείς να κάνουμε ένα mainstreaming ε, σε σχέση με τα δικαιώματα ε, των, ε, των ηθαγενών στα πλαίσια της καθημερινής μας μονομερούς και πολύπλευρης επίσης ή πολυμερούς δράσης σε επίπεδο ε, μονομερές προσπαθούμε να συμμετέχουμε στις διακυβερνητικές συναντήσεις των Ηνωμένων Εθνών είτε στην ετήσια συνάντηση στη Νέα Υόρκη είτε στη συνάντηση του Συμβουλίου στη Γενέβη. Υποστηρίζουμε τις εργασίες των Ταμείων των Ηνωμένων Εθνών στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως επίσης και στηρίζουμε και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για να προωθήσει τα δικαιώματα τα εργασιακά των ε, ηθαγενών και των φυλών που τους αποτελούν. Δίνουμε μεγάλη σημασία στις ειδικέ διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών στη συγκεκριμένη περίπτωση και ιδιαίτερα στις εργασίες του καθηγητή Αλάγια που είναι υπεύθυνο για τα θέματα των ηθαγενών λαών. Βεβαίως το μόνιμο φόρουμ των ε, Ηνωμένων Εθνών για τους ηθαγενείς είναι μια καλή ευκαιρία και πράγματι η όθηση την οποία έδωσε στο θέμα αυτό η απόφαση του 2007 φάνηκε και στη συνάντηση που έγινε τον προηγούμενο μήνα στη Νέα Υόρκη. Υπήρξαν νέε χώρες που συμμετέχουν στην υπογραφή της δήλωσης αυτής, η Νέα Ζηλανδία, οι Ηνωμένε Πολιτείε ενδιαφέρονται και η Κολομβία που συμμετέχει στην προσπάθεια για να συμφωνήσει και αυτή μετά της δηλώσεως. Σε επίπεδο δηλώσεων πάντα, σε αιτήσια βάση γίνεται μία δήλωση του Αρμοδίου Επιτρόπου για Εξωτερικές Υποθέσεις κατά τη διάρκεια με ευκαιρία ε, της ε, ημέρας ε, για τα δικαιώματα των Ιθαγενών λαών που δυστυχώς φέτος είναι η 9η Αυγούστου ξέρετε ότι δεν είναι πολύ εύκολη μέρα λόγω διακοπών. Σε διμερές επίπεδο προσπαθούμε επίσης να συνεργαστούμε με τα γεωγραφικά desk της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καλύψουμε όλες τις χώρες. Αυτός είναι ο πρώτος άξονας ο δεύτερος άξονας είναι να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την Ινδονησία θα υπάρξει ένας νέος διάλογος τον μήνα Ιούνιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προχωράμε λοιπόν σε χώρες ε, με διμερείς διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χώρες ε, για τις οποίες το θέμα των ηθαγενών λαών είναι πάντα χένον. Να υπογραμμίσω επίσης το θέμα και του μέσου που έχουμε στη διάθεσή μας για την ε, δημοκρατία, κάποιες συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως επίσης και των οργανώσεων των υφαγενών. Ένας από τους βασικούς άξονες που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα είναι να χρηματοδοτήσουμε τη συμμετοχή των ΜΚΟ, των Ιθαγενών λαών, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και των συναντήσεων του ΟΗΕ. Αυτό θα έλεγα είναι κάτι το οποίο προσθέτει μία επιπλέον φωνή στις πολυμερείς επαφές. Μπορούμε να επανέλθουμε στις λεπτομέρειες της πολιτικής αυτής αν θέλετε. Εγώ δεν θέλω να αποκλίνω από τον στόχο της ερώτησής σας για την Ινδονησία όμως και γι' αυτό ο συνάδελφος Πέδρο θα ε, συζητήσει τα της Ινδονησίας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κιλ Νίλση μου θέλει και πάλι το λόγο. Oui. Ναι, Πρόεδρε. Γενικός υπήν. Έχω συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία που μετέβη στον ΟΗΕ για αυτούς τους πληθυσμούς. Ε, είναι έκθεση πάρα πολύ άρτια σε σχέση με τις ανταλλαγές απόψεων, τις προτάσεις. Αλλά μία παρατήρηση μόνο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι κάτι που ελέγχθη ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των αντιπροσωπιών στις διάφορες χώρες να ενημερώνεται για τους πληθυσμούς αυτούς. Και είπε ο αντιπρόσωπος στη Νέα Υόρκη ότι πολλές φορές έχουμε την τάση να αρκούμεθα σε αυτές τις επαφές με τους φορείς εδώ στις Βρυξέλλες. Να γίνει κάποια προσπάθεια επομένως πιο άμεση σχέση με τους επιτόπου φορείς όχι μόνο με εκείνους που είναι εδώ στη Βρυξέλλα και έρχονται στο κοινοβούλιο. Αυτό μου είπα να σα διαβάσω. Όντω, έτσι με αντιπροσωπείε γίνεται πιο συστηματικό έργο. Και σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας. Άρα δεν έχετε άλλη ερώτηση. Ωραία. Η Κομισιόν θέλει να συνεχίσει. Να συνεχίσουμε, Πρόεδρε, για την Ινδονησία συγκεκριμένα. Ελπίζω ότι ακρηγόρησα ε, για τις γενικές παρατηρήσεις. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο σας είπα να μας διαβιβάσετε, γιατί όντως υπάρχει προνομική σχέση όσον αφορά τις αντιπροσωπείες και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς για τους ε, αυτόχθονες πληθυσμούς. και ακολουθούν μέσο πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία. Με Καναδά και είπα δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό. Απλώς έχουμε αυτό το χρηματοδοτικό μέσο. Στη Ρωσία όμως υπάρχει και ειδική πολιτική. Ο συνάδελφος Μαρτίνες Βάργκας τώρα θα πάρει τη σκητάλη να σας μιλήσει για την Ινδονησία. Πρόεδρος. Και τώρα ο άλλο πρόεδρο τη Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Καταρχήν, η Κομισιόν ανησυχεί όχι μόνο από τις σειράξεις στην Παπούα μεταξύ της κυβέρνησης και του κινήματος ε, του ανεξάρτητου αλλά και για τα θέματα τα οποία θέσατε εσείς, θέματα γης, ε, αγώνες των ε, τοπικών πολιτικών ομάδων μέσω επικοινωνίας με τη Τζακάρτα. Η Κομισιόν προσπαθεί να παρακολουθεί την κατάσταση εκεί μέσω επισκέψεων, μέσω της συμμετοχής σε συναντήσεις, όπως κάνουμε δηλαδή και με άλλες χώρες, με τη ΣΥΠΑ, την Αυστραλία, την Ζηλανδία, την Ιαπωνία και με πρεσβείες των κρατών μελών για να συζητούμε εκεί επί τόπου στην Τζακάρτα θέματα που αφορούν την Παπουά. Ξέρω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο παρά είναι ευαίσθητο για την κυβέρνηση της συντονισίας οπότε πρέπει να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά όταν θέλουμε να ξεκινούμε διάλογο με την κυβέρνηση στην Ινδονησία για την Παπούα γιατί αμέσως αντιδρούν και θέλουν να σταματήσει οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται για την κατάσταση που επικρατεί στην Παπούα και υπάρχει άρνηση από την ε, κυβέρνηση της Ινδονησίας για, την, το δυναμικό που υπάρχει να ε, επιδεινωθεί η κατάσταση και να κλιμακωθούν οι συγκρούσεις. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά και τα σχέδια της Ινδονησίας για τη μείωση των εκπομπών ανθρακά και βέβαια η παππούα πούμε, αυτό είναι σημαντική. 32 εκατομμύρια εκτάρια καλυμμένα από δάσος έχει η παππούα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων και πρέπει ε, και διοξιδίου του άνθρακα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορεί και τι δεν μπορεί τελικά να κάνει η παππούα. Τώρα, για το θέμα που ρωτήσατε. Ναι, γνωρίζουμε το πρόγραμμα αυτό. Για, την, ε, για το τρόφιμα και την ενέργεια. Θα μπορούσε να καλύψει πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα τμήμα του γενικότερου προγράμματος της κυβέρνησης για την ενίσχυση τέτοιων αγροτικών γεών για την ενίσχυση της επάρκειας σε τρόφιμα και για την ενίσχυση των, των εξαγωγών. Η τελευταία συνάντηση που έγινε με τους ομολόγους του Τζακάρτα ήταν το Μάρτιο με το, με το Υπουργείο Γεωργίας έχοντας ως στόχο καταρχήν να έχουμε πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό και απ' την άλλη να συζητήσουμε κατά πόσο υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, και τρόποι να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της ε, αγροτικής ανάπτυξης στην Παπούα και ταυτόχρονα να, να γίνουν πραγματικότητα και οι δεσμεύσει της χώρας για τη μείωση των εκπομπών αερίων και τα δικαιώματα των αυτοκτόνων στην περιοχή. Και να τονίσω και πάλι ότι όταν μιλούμε για αυτά τα θέματα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση για να μην μας πούν οι αρχές να ξέρετε δεν θέλουμε να το συζητήσουμε όμως το θέμα αυτό και έχουμε και δικαίωμα να μην θέλουμε. Οπότε προσπαθούμε να το θίξουμε με όσο περισσότερο τάκτ και όσο περισσότερη διπλωματία διαθέτουμε. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ακόμα σε φάση προπαρασκευής. Το Υπουργείο Γεωργίας στην Τζακάρτα είναι αυτό που θα πρέπει να δώσει το πράσινο φως. Είναι αυτό που θα πρέπει να ευλογήσει την μετατροπή των γεών. Και ο λόγος για τον οποίο, μάλλον ο λόγος τον οποίο μας δίνει η κυβέρνηση για την όλη καθυστέρηση που υπάρχει για την ε, έγκριση της μετατροπής των ε, γεών, ε, των δασικών γεών σε αγροτική γη, είναι ότι η κυβέρνηση ακόμη χαρτογραφεί την ε, δασική περιοχή στην ε, Παπούα ακριβώς για να αποφύγει τα προστατευμένα δάση από το να γίνουν φυτίες. Το Υπουργείο Δασών μας είπε επίσης ότι ακόμη δεν έχει καθορίσει ε, ποια, θα είναι, θα είναι η γη που θα μετατραπεί σε γη για παραγωγή τροφίμων. Ξέρετε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της Ινδονησίας ήταν στο Όσλο στα πλαίσια της συζήτηση που έγινε για τις κλιματικές αλλαγές και την προηγούμενη εβδομάδα η Ινδονησία υπέγραψε μια συμφωνία με την Νορβηγία μια συμφωνία εταιρική σχέσης για το περιβάλλον και ως ε, τμήμα αυτής της συμφωνίας η κυβέρνηση της Ινδονησίας ξεκίνησε ένα διετές μορατόριο για την ε, δάσωση του συνόλου της χώρας. Οπότε έχοντας και αυτό ως ε, υπόψη μας και τη συμφωνία δηλαδή με την Ορβηγία αλλά και το πρόγραμμα της ε, Παπούα ε, για την, για την, ε, για την τεχνολογία χαμηλού άνθρακα νομίζω ότι αυτό για το επόμενα δύο χρόνια θα σταματήσει. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δύο χρόνια, θα το παρακολουθούμε το θέμα στενά και θα συνεχίσουμε να το συζητούμε με την κυβέρνηση της Ινδονησίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία στην, με την Παπούα για την προστασία του περιβάλλοντος και για το θέμα της, των δασών, η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως χρηματοδοτεί ώστε να μην υπάρξει δάσωση σε αυτό το μεγάλο νησί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Λογοδοσία και Τοπική Πρωτοβουλία για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων ε, το πρόγραμμα RED. Είναι ένα πρόγραμμα που προοικοδοτείται με 100.000 ευρώ που τονίζει κυρίως την συμμετοχή σε τοπικό επίπεδο διαφόρων κοινοτικών ομάδων και στους μηχανισμούς του συγκεκριμένου προγράμματος του RED. Γενικώ, στα πλαίσια της ε, συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδονησίας για τα επόμενα τρία χρόνια από το 2011 έως το 2014 έχουμε συμπεριλάβει και κάποιες νέες προτεραιότητες δηλαδή την κλιματική αλλαγή και στα πλαίσια και της μελλοντική μας συνεργασίας για την ε, κλιματική αλλαγή, όπως είπα για τα επόμενα τρία χρόνια, το θέμα αυτό της ε, αποψηλώσης θα είναι, και, θα είναι αντικείμενο συζητήσεων. Η Παππούα φυσικά θα παραμείνει στην, ε, στις πρώτες θέσεις των θεμάτων προς Επίσης, έχουμε την πρώτη PCA συμφωνία με, την, με χώρα της ε, Νότιο-Ανατολικής Ασίας και αυτό έχει θέσει της διμερείς μας σχέσεις σε πολύ πιο επικοδομητικό και θετικό επίπεδο. Αυτή λοιπόν η συμφωνία προβλέπει συζητήσεις και συνεργασία στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όπως είπε και ο συνάδελφος λίγο πριν, στο τέλος του μήνα θα γίνει η πρώτη συνάντηση για τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Τζακάρτα. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε όχι μόνο θέματα που ήδη είναι στην προσυμπεφωνημένη μερίστη διάταξη, αλλά να μπορέσουμε να θίξουμε και θέματα όπως αυτό εδώ, στο περιθώριο ίσως της συνάντησης αυτής. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Euh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας, η οποία ήταν ε, πλήρης και Αισθάνομαι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτήν. Ο Πρόεδρος, αλλά να ευχαριστήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ξαναδώσουμε πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε το τέλος της εποχής της απερίμωσης των δασών. Και είναι πάρα πολύ σημαντική συνεργασία με δύο χώρες γι' αυτό. Οπότε, κύριε Αντρικένε, κύριε Νίλσεν, σας ευχαριστούμε και εσάς. Πρόκειται όμω, κυρία Κυρινή, να συντάξει μια έκθεση όσον αφορά τη συμμετοχή τη ε, σε αυτή την ε, αντιπροσωπεία που μετέβει στον ΟΗΕ για την ε, διάσκεψη για του θαγενεί πληθυσμού. 11 η ώρα. Έχουμε άλλο θέμα και έτσι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την έκθεση Μάρτιν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εμπορικές συμφωνίες διότι δεν μπορεί να παραστεί επομένως το θέμα αυτό, το υπαριθμό 7 στη μεσή διάταξη αναβάλλεται. Αλλά τέλος πάντων μπορέσαμε να συζητήσουμε για τους ηθαγενείς. Ε, νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Οπότε και προχωρούμε. Στην ακρόαση τη σημερινή που είναι τα δυο μας στην Κεντρική Ασία. Έχουμε πάρα πολλοί εμπειρούς συναδέλφους που έλαβαν ε, μέρος αυτήν την προσωπία και εγώ ήμουν αναπληρώτρια εκεί. Πρόκειται για μια χρονιά που είχε αφιερωθεί στην στρατηγική ε, και την αναθεώρησή τη όσον αφορά τα δικαιώματα στην κεντρική Ασία. Υπήρχαν διαφορετικέ απόψει σε σχέση με το πόσο απέδωσε η στρατηγική μέχρι σήμερα. Οπότε και σήμερα πρόκειται να συζητήσουμε με τους πόλεις μέγεθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα έχουμε επίσης και κάποιους ε, ειδικού από την Κεντρική Ασία. Με την Απροντεύ έχουμε συνδιοργανώσει αυτήν την ε, ακρόαση. Πρόκειται για φορέα ε, που διαπνέεται από εθνικές αρχές. Εγώ, ξέρετε, μαθαίνω Ρώσικα και με μεγάλη μου χαρά θα σας ακούσω να μιλάτε στη γλώσσα αυτή. Για τις εισηγήσεις σας έχετε 10 λεπτά για αυτούς. Παρακολουθούμε αυτά τα όρια γιατί θα πρέπει να γίνει μετασυζήτηση με τους ε, βουλευτές. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και ο κύριος Βαντινή είναι ο πρώτος ε, ομιλητής μας από το Καζακστάν που ασχολείται με θέματα ε, Κεντρικής Ασίας. Ευχαριστώ που δεν αυτή την ευκαιρία κάνω αυτή την εισήγηση και θα ξεκινήσω με μια σύντομη περιγραφή του Καζακστάν για το τι γίνεται εκεί με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχω μια τέταρτη έκθεση και ένα ε, σύστημα ε, μητρώου και όποιο θέλει μπορεί να βρει το κείμενο στην είσοδο τη ε, αιθούσης. Οπότε να σας πω ότι γίνεται όσον αφορά την αστιφιλία στο Καζακστάν, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για μια δουλειά που αφορά την, την ιστορική μετανάστευση και, τις, τη μετανάστευση γενικά, τις ροές που είναι πάρα πολύ έντονες το 2007 οι περισσότεροι μένανε στην ε, Ήπεθρο ε, πάρα πολύ χαμηλό το βιωτικό επίπεδο και δεν υπήρχαν δουλειές και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί πήγανε στις ε, πόλεις Άλμα Άτα ή σε άλλες πόλεις του κεντρικού Καζακστάν για να δουλέψουν στις ε, οικοδομές και σε άλλους ε, τομείς της οικονομίας και έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους της ε, Υπέθρου οι οποίοι πήγανε στις πόλεις. Αυτό έγινε από το 2003 με το 2007. Μήπως μπορείτε να μιλήσετε πιο αργά, λέει η Πρόεδρος. Πάνω από ένα εκατομμύριο, λέει ο εισηγητή. Κάτοικοι τη Υπέθρου ε, μετανάστευσαν εσωτερικά για αυτήν την πενταετία. Πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό. Πολλές φορές είναι αδήλωτοι. Δηλαδή στην πόλη παραμείνουν δεν δηλώνονται στο σχετικό μητρό, οπότε υπάρχει πρόβλημα άσκησης των δικαιωμάτων τους. Σύμφωνα με το νόμο της χώρας, υποχρεούνται να δηλωθούν εάν αλλάξουν τόπο κατοικίας. Επίση, εάν ε, έστω και προσωρινά την κατοικία πάνω από τρεις και αυτό πρέπει να το δηλώσουν. Και βέβαια αυτό διέπεται από κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις και έχει να κάνει και με την ενοικίαση σε κάποιο σπίτι, κάποιο διαμέρισμα. Οπότε γίνεται και έλεγχο του κατά πόσο κρίνονται κάποιε προδιαγραφέ ασφάλεια κλπ. τη ανοικοδόμηση αυτού του τόπου κατοικία. Οπότε υπάρχουν και κάποιε κυρώσει αυστηρέ για αυτού οι οποίοι δεν έχουν δηλωθεί. Αν και άλλαξαν τόπο κατοικία. Παρά την φιλελευθερωποίηση της δεκαετίας του 90, τη μείωση της γραφειοκρατίας από το 2005 και μετά αυτό το σύστημα του αρχείου μπορώ να πούμε ότι ήταν κληροδότημα της Σοβιτικής Ένωσης. Βέβαια, δεν υπάρχουν τόσοι περιορισμοί μετακίνηση όπω στην εποχή τη Σοβιετική Ένωση δεν αποτελεί μέσω ελέγχου της ιστορικής μετανάστευσης. Όμως, ακόμα υπάρχουν πολλές φωνές αντίθετες σε σχέση με αυτό το σύστημα. Ε, κυρίως είχαμε πρόβλημα με το, με το Κυργιστάν πέρσι, αλλά και όλα αυτά λόγω της οικονομικής ύφεσης ε, γίνανε πιο έντονα. Αυτό το σύστημα πάνω του να δηλώνει και αυτόν τον τόπο κατοικίας του έχει να κάνει με την άσκηση των κοινωνικών και άλλων δικαιωμάτων όμως θα πρέπει να προσάγονται αποδείξεις για τον τόπο κατοικίας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει αυτός που δηλώνεται να έχει κάποια δήλωση ε, ιδιοκτησίας κάποιου ακινήτου ή δήλωση από μέλη της οικογένειας του των φιλοξενούν. κοινωνικά επιδόματα, υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ακόμα και η πρόβαση στη δικαιοσύνη ρυθμίζεται από αυτό το σύστημα του ληξιαρχείου, τέλος πάντων του, του, του δημοσίου μητρώου. Οπότε οι άστεγοι και άλλοι κοινωνικά ευάλωτοι θα πρέπει να αποδείξουν που μένουν, θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν δηλωθεί για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίε κοινωνικής πρόνοιας και στα επιδόματα. Ε, και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι δεν, έχουν, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση λόγω του ότι είναι ακριβές υπηρεσίες των ιδιωτικών φορέων. ούτε υπάρχει πρόβλεψη. Πρέπει να τα λέτε πιο σιγά, λέει ο πρόεδρος. Οπότε υπάρχει να προσφέρουν στην ε, δικαιοσύνη, δεν μπορούν να προσφέρουν στην δικαιοσύνη αν δεν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν δηλώσει την τοποκατοικία τους. Τώρα αυτά ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένα για να δούμε τώρα κάπως, κάπως ευρύτερα ζητήματα. Ε, αυτά τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνική αρρωγή. Βέβαια και αυτά τα προγράμματα σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας θα επιληθούν αυτόματα λέγαμε τα κοινωνικά θέματα γιατί θα υπάρξουν κονδύλια. Όμως αυτό δεν ισχύει αναγκαστικά δείχνει η εμπειρία. Η κυβέρνηση προβλέπει κάποια κοινωνικά επιδόματα, όμως δεν μπορούν να καλυφθούν κάποιες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, περισσότερη διαφάνεια στο σύστημα δικαιοσύνης και προσβασιμότητας από κάποιες κοινωνικές ομάδες, αλλά όχι για όλους. Είμαι ειδικό στα μετανάστευση και είμαι στη να ξέρω ότι η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται όπως θα έπρεπε. Και αυτές τις νέες προκλήσεις δεν τις αντιμετωπίζει. Παράδειγμα, στο Καζακστάν έρχονται σαν μετανάστες ένα εκατομμύριο άνθρωποι από Ουσβεγιστάν, Κυργιστάν, δύο από τις όμορες κεντροασιατικέ χώρε. Πέραν της εσωτερικής μετανάστευση που προαναφέραμε. Είχαμε μια ειδική επιτροπή για την μετανάστευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας αλλά κυρίως ασχολούνται με τον επαναπατρισμό των Καζάκων που κατοικούν στο εξωτερικό. ξεκίνησε το πρώτο αυτό το δεκαετία του και συνεχίζεται, όμως έχουμε και άλλες μεταναστεύσεις που γίνονται όλο ένα και πιο σημαντικές και δεν καλύπτονται από αυτή την Επιτροπή. Γιατί? Διότι είναι ευκολότερο να εισπράττονται τα κονδύλια για τον επαναπατρισμό και να μην ασχολείται αυτή η Επιτροπή με τα δικαιώματα των οικονομικών μεταναστών. Δύο φορές έκανα σχετικό διάβημα στο κοινοβούλιο μας, αλλά ακόμα περιμένω τα αποτελέσματα. Και θα κλείσουμε το εξής. Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, περισσότερη στα στην κοινωνική πολιτική και αυτό θα φέρει σταθερότητα στην περιοχή γιατί υπάρχει φτώχεια, δεν, δεν υπάρχουν τα κοινωνικά δικαιώματα και αυτό είναι κάτι το οποίο αντανακλάται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Θα πρέπει επομένω η κυβέρνηση να εξασφαλίσει το ότι οι ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε να μπορούν να έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα τα επιδόματα τη κοινωνική πρόνοια θα πρέπει να, να, να, να είναι προσβάσιμα από όλο τον κόσμο. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε και στα πλαίσια τη στατίκη τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε και τα προγράμματα τεχνική αρρωγή με την Κεντρική Ασία. Οπότε σα προτείνουμε να διερευνηθεί το Πώς μπορούμε να τα καλύψουμε αυτά τα κοινωνικά θέματα, να τα κάνουμε προτεραιότητα σε αυτόν τον πολιτικό διάλογο υψηλού επίπεδου. Στα πλαίσια πάντα της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία. Και σε αυτό το διάλογο να εμπλέκονται τα συναρμόδια Υπουργεία. Απασχόληση κοινωνικής πρόνοια παιδεία, υγεία. Το ίδιο να ισχύει τα προγράμματα τεχνικής αρρωγή και να βοηθήσουμε τους ευάλωτους όπως τους ε, οικονομικούς μετανάστες, τα παιδιά, τους άστεγους. Και τα θέματα γενικής πολιτικής μπορούμε να τα διεκπαιρεώσουμε στα πλαίσια των ενωσιακών πρωτοβουλειών. και να δούμε και τι θα γίνει για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη αυτών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Και εγώ ευχαριστώ. Ακό, αργότερα θα έρθει να μας μιλήσει η κυρία Γέγκλε, η, της οποίας η Επιτροπή επισκέφτηκε το Καζακστάν πρόσφατα. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γιακούποβα, η οποία είναι πρόεδρος στο Κυργιστάν μιας τράπεζας νομικών υπηρεσιών. Καλημέρα σας. Uh, uh, Μετά από αυτά που ακούστηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές είναι εύκολο για μένα να περιγράψω την κατάσταση. Νομίζω ότι ο νόμος ε, γενικά και η επιβολή του νόμου και ο σεβασμός της νομικής τάξης είναι κάτι το οποίο ισχύει σε όλο τον κόσμο ή πρέπει να ισχύει σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα πλαίσια. And maybe the example and the last events in our country η κατάσταση στη χώρα μου νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει μια καλή εικόνα για το πώς ε, έχουν τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή. Βασικός στόχος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Κεντρική Ασία είναι η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή. Ε, it's excluded from public life and... Uh, Κάποιοι οι οποίοι ίσως να μην είναι επίσημα καταγεγραμμένοι. In various levels. According our research in Kyrgyzstan, there it's about 20% uh, of uh, local population. Από ό,τι καταλαβαίνουμε στο Κυργιστάν, το 20% του πληθυσμού αποκλείονται από τη δημόσια ζωή. From... Την παιδεία και την ιατρική και κοινωνική βοήθεια. Uh, uh, Το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί σήμερα δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να είναι αποτελεσματική στις παρεμβάσεις της. Έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου η απουσία είναι σαφής, σε πολλές περιπτώσεις και στην νοσοκομιακή περίθελψη και στην παιδεία. The Propiska system is one of the instruments of manipulation of results of election. And all these factors were played, played very negative role Όλα αυτά έχουν παίξει πάρα πολύ αρνητικό ρόλο. Η περιθωριοποίηση τμήματων του πληθυσμού είναι σαφής. Και ακριβώς αυτοί οι περιθωριοποιημένοι πολίτες χρησιμοποιήθηκαν από τα διάφορα πολιτικά κόμματα σε αυτό που ονομάζουμε Επανάσταση του 2005 και στα γεγονότα του μηνός Απριλίου του 2010. Μετά τον Απρίλιο του 2010, όταν έφυγε ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Μπακίευ... σκοτώθηκαν 100 πολίτες και ξεκίνησε η τοπική κυβέρνηση προετοιμασίες ε, για ένα δημοψήφισμα και εκλογές για το Κοινοβούλιο και την Προεδρία. Υπάρχει όμως ε, μια δυσκολία σχετικά με την ερμηνεία των ρυθμίσεων του συντάγματος και δεν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση και να επικρατήσει το κράτος δικαίου γενικότερα στη χώρα μας. Σύμφωνα με την τελευταία διατύπωση της συνταγματική, τα δικαστήρια εξαρτώνται uh, εξαρτώνται από το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση. είναι δύσκολο να επικρατήσει το κράτος δικαίου. Στα πλαίσια της προετοιμασίας για τις εκλογές και το δημοψήφισμα, πολλά πολιτικά κόμματα προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα της Πραπίσκα για να παρέμβουν αρνητικά και να στρεβλώσουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Παπρίσκα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση με τη μέθοδο αυτή, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αυτό σε όλη την Κεντρική Ασία. Συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για μας αν βάλουμε στην ημερήσια διάταξη ε, των συναντήσεων υψηλού επίπεδου πιο συγκεκριμένα θέματα όπως το παπίσκα. Αυτό θα είναι κάτι το χρήσιμο then I think it would be useful if we can strengthening the θέμα είναι interagencies and and interagencies and regional and international cooperation on Μήπως μπορούμε να ενισχύσουμε την συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές δομές και στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Πριν έρθω εδώ, συναντήθηκα με κάποιες αμερικανικές υπηρεσίες και είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει το σύστημα παπίσκα στο Κυργιστάν. Υπήρξαν θερμότατες συζητήσεις και στα πλαίσια των προγραμμάτων του Ταμείου Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών και στα πλαίσια των προγραμμάτων του ΟΑΣΕ για να αλλάξει η νομοθεσία στο Κυργιστάν και να γίνει πιο στενή συνεργασία με την κυβέρνηση για την αλλαγή του συστήματος Παπίσκαν. Καλό θα είναι λοιπόν όλες οι επαφές που θα γίνουν να μην αγνοήσουν ε, το πρόγραμμα αυτό και σε διεθνές επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο. η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνει την προσοχή της περισσότερο στη συνεργασία με τις κυβερνητικές δομές. Αλλά τα παραδείγματα που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι δυστυχώς όταν γίνονται πολιτικές αλλαγές σε πολλές περιπτώσεις αλλάζει το πολιτικό προσωπικό. και πολλοί εκπαιδευμένοι υπάλληλοι χάνουν τη θέση τους και δεν μπορούν να προσφέρουν. Όταν αλλάζει η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται με την τεχνογνωσία που έχει το προηγούμενο πολιτικό προσωπικό και θα πρέπει στο πρόγραμμά σας γύρω από τον τομέα αυτό να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Of Θα πρέπει να υπάρξει και ένα τεχνικό πρόγραμμα, όπως είπε και ο Βαντίμ, ένα πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για τις κυβερνητικές υπηρεσίες να υπάρξει ένα πρόγραμμα πληροφορικής για να αλλάξει το σύστημα καταγραφής παπίσκα. Uh, for providing, uh, you know, experts from European countries, from countries or uh, υπάρχουν πολλές χώρες της περιοχής, υπάρχουν πολλές χώρες ακόμα και μέχρι τη Βαλτική που έχουν αλλάξει το σύστημα παπίσκα στη χώρα τους και στις οποίες χώρες μάλλον έχει δοθεί τεχνική βοήθεια για να προχωρήσουν στις αλλαγές της Παπίσκα. Εμείς δεν έχουμε εμπειρογνώμονες στην κυβέρνησή μας για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει το σύστημα. Ευχαριστώ. Παπίσκα. Εγώ ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον τρίτο μιλητή, την κυρία Νιάσοβα. Είναι πρόεδρος του Φόρουμ για, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δραστηριοποιείται και στο Ουσβεκιστάν και στη Γερμανία. Ευχαριστώ ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Ουσμπικιστάν είμαι. Έχω δύο χρόνια που έχω φύγει από το Ουσμπικιστάν μετά από μια υπόθεση στο δικαστήριο. Τώρα ζω στο Βερολίνο. Ε, πολλοί συνάδελφοί μου είναι στην ε, φυλακή τώρα για τη δραστηριότητά τους ε, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο Ουσμπεκιστάν η Σοβιετική εποχή άφησε αυτή την υποχρεωτική καταχώρηση καταγραφή που ονομάζεται Παπίσκα. Ή το σύστημα αυτό επιτρέπει στο κράτος όχι μόνο να καταχωρεί το, το τόπο διαμονής των πολιτών, αλλά θέτει σε μεγάλο έλεγχο τις δραστηριότητες και την μεταφορά τους. Όλοι πρέπει να έχουν ένα, μια σφραγίδα στο διαβατήριό τους. Και χωρίς αυτό οι πολίτες δεν έχουν δικαίωμα να ε, εγκαθίστανται σε ένα συγκεκριμένο μέρος ούτε να φύγουν από τη χώρα. Οπότε χάνουν πολλά άλλα δικαιώματα όπως ε, στέγαση, ε, εργασία, εκπαίδευση, δικαίωμα να παντρευτούν. Το 2009 οι τοπικές ομάδες έκαναν μια έρευνα για την ελευθερία κίνησης και με βάση την έρευνα που έγινε υπήρξε μία έκθεση καθώς και συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι, εσωτερικός, με, ε, οι άνθρωποι που έχουν μεταφερθεί σε, άλλο, σε άλλα μέρη εκτοπισμένοι και που θέλουν να ε, μετακομίσουν και να ζήσουν αλλού ε, υπόκεινται σε ε, πολλούς περιορισμούς και νιώθουν σαν ξένοι στη χώρα τους στην Τασκένδη υπάρχει πάρα πολύ δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, ειδικά σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των πολιτών και την ελευθερία κίνησης. Οι πολίτε από άλλε περιφέρειες της, ε, του Ουσμπικιστάν που φτάνουν στην Τασκένδη ε, πρέπει να καταγραφούν ε, για την κατοικία τους και οι κανόνες για τη διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ περίπλοκοι, δύσκολοι και χρειάζονται και χρήμα και χρόνο οι Ουσμπέκοι που έρχονται στην ε, πρωτεύουσα πρέπει σε μέσα σε τρει μέρε από τη μέρα που θα φτάσουν να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να καταχωρηθούν στο Υπουργείο Ιστορικών. Όλοι αυτοί πρέπει να έχουν ε, αποσύρει τα, χρήματα, τα, ε, τα έγγραφά τους από, την προηγούμενη, από το προηγούμενο μέρος κατοικίας τους. οι αρχές εξασφαλίζουν την ασφάλεια όλων αυτών και ή αν κάποιο θέλει να πάει να δουλέψει για λίγο ή για σπουδέ, πρέπει να πάρει άδεια μικρής διάρκεια. Και αυτό πάλι πρέπει να γίνει μέσα σε τρει μέρε που θα φτάσει στο σημείο που θα σπουδάσει ή θα δουλέψει. Για να πάρει αυτή την ε, άδεια. Καθορίζεται το αντίτιμο που πρέπει να πληρώσει και η πληρωμή δεν έχει όριο. Οι πολίτες μπορούν, πρέπει πολλές φορές να χρησιμοποιήσουν ε, και να δωροδοκίσουν ε, υπαλλήλου για να πάρουν τα έγγραφα που χρειάζονται. Το Υπουργείο Ιστορικών συντονίζει το όλο σύστημα παροχής ε, έκδοσης διαβατηρίων σε συνεργασία βέβαια και με την τροχέα, τις άλλες ερευνητικές υπηρεσίε ώστε να βρούνε ποια είναι τα, ποιοι είναι οι πολίτες που έχουν ε, ε, διαβατήρια και δεν έχουν άδειε ε, διαμονής. Οπότε μόλις βρεθούν αυτοί ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές για την παρανομία που έχουν κάνει αυτοί οι πολίτες. αυτοί που δεν μπορούν να λάβουν ε, τελικά ε, άδεια παραμονή δεν μπορούν να απασχοληθούν σε καμία επιχείρηση, σε κανέναν οργανισμό που βρίσκεται σε αυτή την περιοχή. Και σύμφωνα με τους κανόνες πρέπει να φύγουν μέσα σε 7 ημέρες. Αν δεν φύγουν μπορεί κάποιος να απελαθεί από τις αρχές από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό αφορά και περιορισμούς ε, και για τις άδειε ε, ε, παραμονής και στην Τασκένδη και σε άλλες περιοχές. Οπότε ο περιορισμός αυτό σημαίνει και παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και, δείχνει ότι υπάρχουν και μεγάλα, πολλές περιπτώσεις δωροδοκίας σε διάφορες υπηρεσίες. Στην Τασκένδη απαγορεύεται αν δεν έχει κάνει την άδεια να αγοράσει ε, την κατοικία του. Σε μια συνέντευξη με έναν πολίτη από κάποια άλλη περιοχή ε, μου είπαν ότι, είπαν ότι δεν, ένα, για 12 χρόνια δεν ήμουν καταχωρημένος επειδή δεν ζούσα στην περιοχή εκεί και μόνο όταν με δωροδόκησα τους υπαλλήλους μπόρεσα να πάρω την άδεια και να καταγραφώ. Πολλοί έχουν καταφέρει να βρούνε βέβαια δουλειά χωρίς την, χωρίς την άδεια. Η κατάσταση όμως αυτή πραγματικά είναι γεμάτη κινδύνους γιατί οι τοπικές αρχές κάνουν συχνά ελέγχους ώστε να συλλάβουν άτομα χωρίς άδεια παραμονής και που δεν είναι καταχωρημένα. Και πολλοί πρέπει να δωροδοκίσουν ε, τους αστυνομικού ή τους ε, υπαλλήλου τη τοπικής αστυνομία για να είναι υπό την προστασία τους. Οι πολίτε που φτάνουν στην πρωτεύουσα από την περιφέρεια λένε ότι συνεχώ τους ζητούσαν ε, να δωροδοκίσουν για να μπορέσουν να ζήσουν και να εργαστούν στην πρωτεύουσα. Μία κυρία που δουλεύει στην Τασκένδη στην συνέντευξη είπε ότι είχα διακοπές και σε εκείνες τις μέρες άρχισαν, έγιναν ε, έλεγχοι από την αστυνομία και εγώ ε, μου απαγόρευσε η αστυνομία να βγω έξω μαζί με τα παιδιά μου. Έπρεπε να πληρώσω 8 δολάρια στο αντίστοιχο τοπικό νόμισμα για να μπορώ να βγαίνω κάθε τέλος του μήνα από το σπίτι μου αστυνομία ελέγχει τα διαβατήρια και έτσι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες ε, να δολοδοκίσεις κάποιον για να να, για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά σου. Στην Τασκένδη έχω δει πολλές φορές ε, αστυνόμους να σταματάνε κόσμο στο δρόμο να, ελέγχει, τα, να ελέγχουν τα διαβατηριά του, μόνο και μόνο γιατί δεν μοιάζουν με πολίτες της πρωτεύουσα. Πολλές φορές οι πολίτες λένε ότι με ανάγκασε κάποιος να δουλέψω στο σπίτι του ή στο σπίτι φίλων του κάνοντας διάφορες δουλειέ και ε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας υπάρχει πάνω από ένα εκατομμύριο ατόμων εκτοπισμένων από την περιφέρεια που έχουν πάει για δουλειά στην, ε, στην ε, πρωτεύουσα. Επίσης, ε, το σύστημα της ε, καταχώρησης ε, δικαιολογείται από την ανάγκη που υπάρχει να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία και ο εξτρεμισμός. Πρακτικά όμως το σύστημα αυτό καταχώρησης είναι ένας παράδεισος διαφθοράς. Οι μόνιμοι, οι μόνιμοι κάτοικοι ορίζονται από την απόφαση που βγάζει η Ειδική Επιτροπή Καταχώρησης. Ε, η διαφθορά και το ποσό φτάνει της διαφθοράς των ευρωπαϊκών φτάνει και τα 5.000 δολάρια. Η Επιτροπή αυτή θυμίζει μια σταλινιστική περίοδο ε, και το Υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνει μέσα σε δύο μέρες ε, τα έγγραφα τα οποία πρέπει να στείλει στην αρμόδια αρχή και μέσα σε δέκα μέρες η αρμόδια αρχή πρέπει να δώσει την απάντησή της για το κατά πόσο αυτός ο ετών είναι αξιόπιστος. Αλλά εξακολουθεί να είναι ασαφές πώς ακριβώς ε, ε, ορίζει την αξιοπιστία ενός ατόμου αυτή η Επιτροπή. Όλοι όσοι ρωτήσαμε είναι άνθρωποι από την, ε, κυβέρ... από την Ήπεθρο ε, ε, που ήρθαν στην πρωτεύουσα να, πάρουν, να βρουν δουλειά και φυσικά κανένας δεν είχε τα... το αντίστοιχα χρήματα για να πάρει την άδεια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θεωρούνται ότι έχουν παραβιάσει το καθεστώς για, για τα διαβατήρια και τίθενται υποκράτηση και σε κέντρα τα οποία έχουν ως στόχο να να κρατήσουν εκεί τους ανθρώπους αυτούς γιατί τους βρήκανε χωρί τα απαραίτητα έγγραφα ή το διαβατήριο. Ένας ακτιβιστής μπήκε σε αυτό το, το κέντρο για 15 μέρες και μα είπε μετά ότι οι υπάλληλοι αυτού του κέντρου ε, εξευτελίζουν τους κρατούμενους, τους προσβάλλουν, τους χτυπούν, ε, τους ζητούν χρήματα και η αστυνομία δεν ξεκαθαρίζει φυσικά ποτέ την κατάσταση. παρόλο που μπορεί να έχουν τα έγγραφα με την ταυτότητά του, εξακολουθούν να κρατούν τους ανθρώπους αυτούς μέχρι να τους πληρώσουν, μέχρι να τους δώσουν χρήματα για να φύγουν. Άλλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ουσμπέκων συμβαίνουν λόγω του συστήματος για την θεώρηση εξόδου. Πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν ε, πρέπει να πάρουν άδεια που ισχύει μόνο για δύο χρόνια. Η άδεια αυτή ε, εκδίδεται ως αυτοκόλλητο που μπαίνει στο διαβατήριο του ετούντα, όπως η θεώρηση εισόδου. Αυτή ονομάζεται θεώρηση εξόδου πάλι από τη Σοβιετική εποχή έχει κατάλοιπο. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος αυτός να ταξιδέψει στις χώρες αυτές Οι χώρες CIC ε, δεν χρειάζονται θεώρηση για να περάσει κανεί. Αλλά χώρε όπω η Ρωσία και το Καζακστάν έχουν ε, υπογράψει με το Ουσμπεκιστάν συμφωνία που λέει ότι απαγορεύεται οι Ουσμπέκοι να φύγουν από τι χώρε αυτέ για χώρε άλλε εάν δεν έχουν θεώρηση εξόδου. Οι πολίτες του Ουσμπεκιστάν που θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες πρέπει να πάνε στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών στην περιοχή που μένουν, να συμπληρώσουν μια αίτηση και να υποβάλουν το διαβατήριό τους. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ε, πολιτών που αντιμετωπίζουν τέτοια διάκριση σε ό,τι αφορά το, τα ταξίδια, οι δημοσιογράφοι, οι ε, εκτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάποιες θρησκευτικέ κοινότητες και τα μέλη τους. Τον Ιούνιο του 2009 ο Πρόεδρος εξέδωσε ένα διάταγμα για την εισαγωγή νέου διαβατηρίου βιομετρικού για τους ε, πολίτες με τα προσωπικά τους δεδομένα. Δυστυχώς όμως το διάταγμα αφήνει το σύστημα καταχώρησης απαράλλαχτο. Καθώ επίσης και τις συνθήκες για να μπορεί να μπει ή να βγει κανείς από τη χώρα. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν την εμπειρία τριών χωρών για την ε, σοβιετική κληρονομιά που έμεινε και πώς χρησιμοποιείται και πώς ε, ε, την καταχρώνται οι αρχές και παραβιάζουν τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Τώρα η Κομισιόν ας μπει στη συζήτηση. Έχουμε εδώ από τη Γενική Διεύθυνση ΡΕΛΕΚΣ τον κύριο Άλβαρες Μαλδονάδο και στην αρχή είπα ότι φέτος είναι το έτο ε, όπου θα αναθεωρηθεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωση για τις χώρες της Κεντρικής Ασία. Οπότε, κύριε Μαλτονάδο, τι έχετε να απαντήσετε. Και επίσης μπορείτε να σχολιάσετε την κατάσταση των ε, ακτιβιστών ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Εντάξει, δεν είναι το αντικείμενο αυτή της συγκεκριμένης συζήτησης, αλλά Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο θέμα και η κυρία Νιάσοβα το ανέφερε ότι πολλοί από τους συναδέλφους της ε, αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένοι. Οπότε ας μην το ξεχνούμε αυτό. Έχετε το λόγο λοιπόν. Thank you, Well, I was prepared... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ήμουν έτοιμος να σχολιάσω αυτά που είπε ο προηγούμενος ή η προηγούμενη συνάδελφος, τέλος Μπα και μπορώ να το κάνω. Καθώ τον θα έτσι πάρα πολύ. Σύντομο, ε, όπω είπατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η στρατηγική τη Ένωση για την Κεντρική Ασία εγκρίθηκε στο Συμβούλιο το 2007. Και είναι θέμα αξιών. Περί αυτού πρόκειται. Πάρα πολύ σημαντικό. Οι αξίε που τα στα κλπ. Και γι' αυτό είναι στην καρδιά αυτού του οράματο, διότι έχουμε πιστεί ω Ευρωπαίοι ότι με αυτόν τον τρόπο καλύτερα θα μπορέσουμε να ε, ρυθμίσουμε τα θέματα του, του, του, του πληθυσμού κλπ. Επίση, είμαι θα ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε όσο γίνεται περισσότερη ευημερία του πληθυσμού στην Κεντρική Ασία, αλλά θα βοηθήσουμε και την ε, ανάπτυξη όλων των χωρών στην περιοχή. Αυτό φαίνεται αυτονόητο, αλλά δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε ότι αυτό είναι η καρδιά, το επίκεντρο της στρατηγικής. Αξίες, αξίες. Πώς όλα αυτά τώρα υλοποιούνται. Έχουμε δύο άξονες. Πρώτα-πρώτα πολιτικός διάλογος, ο οποίος έχει διευρυνθεί την τελευταία τριετία πάρα πολύ. Οπότε, πριν είχαμε σε σε επίπεδο υπουργικό Τώρα έχουμε δύο υπουργικές συναντήσεις ετησίως και συζητούνται τα πάντα, όλα. Και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξέρετε ότι είμαστε η μόνη ομάδα στον κόσμο που έχει πέντε συναντήσεις διαλόγου τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις χώρες αυτές. Αυτό μην το ξεχνάτε. Ούτε οι άλλε ούτω οι μεγάλε δυνάμει κάνουν τέτοια πράγματα. Διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βέβαια, αυτό είναι χρονοβόρο. Θέλει υπομονή, δεν λύνονται τα θέματα από τη μια μέρα στην άλλη. Όμω έχουμε ολοκληρώσει δύο γύρου επαφών. Έγινε με θα γίνει τώρα για Τουρκμενιστάν και για τις άλλες δύο χώρες αργότερα. Αυτό δείχνει ότι είναι σταθερή η προσήλωσή μας σε αυτά τα θέματα και σας ε, διαβεβαιώ ότι όλα τα ζητήματα τίθενται σε αυτές τις επαφές. Παπίσκα, προπίσκα το σύστημα αυτό τέλος πάντων οι, όλες αυτές οι λαθροχειρίες, οι καταχρήσεις όλα αυτά με συγκεκριμένο τρόπο τίθενται επί της τραπέζης. Σας διαβεβαιώ Όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι εδώ εκ δεξιών, όλα αυτά με συγκεκριμένο τρόπο τα θέσαμε. Επίση, μετά από τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε και το θέμα του κράτου δικαίου. Είναι μια πρωτοβουλία, μια κοινή προσπάθεια από τι κυβερνήσει, τι κεντρεσιατικέ, αλλά και από την Ένωση. Ούτω ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά το να υπάρχει κράτο δικαίου στην, στην κεντρική Ασία. Άρα, εκεί εστιάζουμε την προσοχή μα σε κάποια θέματα που για μας φαίνονται αυτονόητα, αλλά μόλις τώρα αρχίζουν να τα καταλαβαίνουν στην Κεντρική Ασία. Δηλαδή, ας πούμε, οι ανεξαρτητές δικαιοσύνης, η προσβασιμότητα στη δικαιοσύνη, τι, τι πλέον εκτίματα προσφέρουν, καλύτερη κατάρτιση εκπαίδευση δικαστών. Οπότε όλοι αυτοί στην Κεντρική Ασία τώρα τα καταλαβαίνουν καλύτερα αυτά τα θέματα, βέβαια αυτό θέλει χρόνο, Αλλά πριν ε, προχωρήσουμε στις λεπτομέρειες, για να δούμε πρώτα αυτό για την προπίσκα και το μητρό, θα πρέπει να γίνει εδώ μια διαφοροποίηση μεταξύ, μεταξύ χρήσης ε, αυτού του μητρώου σαν μέσο καταστολής και ελέγχου. Και από την άλλη μεριά υπάρχει η τεχνοκρατική άποψη του ζητήματος που βέβαια επιδέχεται επίσης κακοδιοίκηση, ε, επιδέχεται μικροφαινόμενα διαφθοράς. Όμως θα πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση. Άρα, σαν κρατική καταστολή χρησιμοποιούμενο το σύστημα, αυτό ήταν πρόβλημα το οποίο συζητήθηκε στον διάλογο ένας της Κεντρικής Και να μην ξεχνούμε ότι τέτοιο σύστημα ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα το, το, το, πρόβλημα δεν είναι η ιδέα, το σύστημα. Το θέμα είναι πώς κανείς χρησιμοποιεί, καλός ή κακός και για ποιο σκοπό το σύστημα. Να αποφύγουμε περιθωριοποίηση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Να αποφύγουμε το σύστημα αυτό να χρησιμοποιείται ή σαν συνέπεια να έχει το να μην μπορεί κανένας να, να, να ωφεληθεί από κάποια επιδόματα, να μην μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη αν δεν έχει εγγραφεί στο Μητρό. Οπότε, για, για το σκοπό της ε, καταστολής, αυτό είναι εις βάρος του κόσμου, αλλά τα προβλήματα για τη δεύτερη εκδοχή είναι ένα πρόβλημα που κληροδοτήθηκε από την προηγούμενη κατάσταση. Και όπως προείπα για τον έλεγχο του λαού αυτό συζητήθηκε στον πολιτικό διάλογο και όσον αφορά τις καταχρήσεις του συστήματος αυτό συζητήθηκε επίσης σε πολιτικό επίπεδο και υπουργικό επίπεδο αλλά όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης ασχοληθήκαμε με το πώς θα εφαρμοστεί το σύστημα και διερμήσαμε διαφορετικές δυνατότητες που προσφέρονται οπότε και τώρα προσπαθούμε όλα αυτά τα προϊόντα να τα εντάξουμε στα προγράμματα, άρα έχουμε την πρωτοβουλία του κράτους δικαίου, έχουμε τα σεμινάρια, τις διασκέψεις, ε, τις συναντήσεις, οπότε και από εκεί προκύπτει ποια είναι τα βασικότερα στοιχεία, ε, τι προτάσεις, τι συστάσεις υπάρχουν για το σύνολο αυτής της γεωγραφικής περιοχής. Και πρόκειται για κοινή προσπάθεια, η μόνη και εκείνων. Έχουν συμμετάσχει αυτές οι πέντε χώρες πάρα πολύ δυναμικά. Ανώτατοι δικαστές ήρθαν και έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Επίσης έχουμε και κάποιες άλλες ε, επαφές ε, διημερείς όπως για το κράτος δικαίου. Διμερείς γιατί θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη η μερικά κάθε χώρα, δεν είναι δυνατόν η ίδια συνταγή να ακολουθείτε για όλους. Να σας πω κάποια παραδείγματα. Στο μέλλον πρόκειται να έχουμε ένα πρόγραμμα 14 εκατομμυρίων για το Κυργιστάν και το κράτος δικαίου. 14 εκατομμύρια, πολλά λεφτά. 25 εκατομμύρια προβλέπεται να διατεθούν για το Ουσμπεκιστάν, πάλι για το κράτος δικαίου. Και την δικαστική μεταρρύθμιση. 25 εκατομμύρια, πολλά λεφτά. 10 εκατομμύρια για το δικαστικό σύστημα για τη δικαιοσύνη στο Καζακστάν. Επομένω, κρίθηκε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωση και να έχουμε δυνατότητα να προοδεύσουμε, να βελτιώσουμε και το σύστημα αυτή τη ε, καταχώρηση στο Μητρό. Γιατί υπάρχουν πολλέ αντιρρήσει, πολλέ αρνητικέ συνέπειε. Αλλά βέβαια εδώ προποτίθεται να υπάρχει και πολιτική βούληση. αυτά τα προγράμματα καλύπτουν πολλούς τομείς και άρα θα πρέπει να τάξουμε για τις προτεραιότητες και να διαλέξουμε. Ας πούμε προσωπικά με καίει το θέμα της εξαρτησίας της δικαιοσύνης. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Θα υπάρχουν και άλλα ζητήματα όπως η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η εκτέλεση των αποφάσεων της εισαγγελίας. Πολύ σημαντικά. Άρα θα πρέπει για κάθε θέμα κανείς να βλέπει ποια προτεραιότητα θα κατησχύει. Και όλα αυτά με τα δεδομένα χρήματα που έχουν στη θέση μας. Τώρα, κοινωνική πρόνοια. Και εδώ έχουμε προγράμματα για όλες τις χώρες. γιατί και εδώ είναι το θέμα του Κυργιστάν και άλλων χωρών της μη πρόσβασης στην κοινωνική πρόνοια γιατί έχουμε και 20 εκατομμύρια που προβλέπονται για το Καζακστάν και 19 στην Κυργισία και 12 για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Οπότε θα πρέπει αυτά τα προγράμματα να τρέξουν Και θα πρέπει οι συνάδελφοι εδώ και δεξιόν μου να έρθουν σε επαφή με τις αντιπροσωπείες σε Κυργιστάν, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν να έρθουν σε επαφή με τις αντιπροσωπείες γιατί αφού λέμε για 10-20 εκατομμύρια υπάρχει πολύ περιθώριο για να κινηθούμε και να μπορέσουμε να δούμε και τι τεχνική αρρωγή θα δοθεί από μέρους μας. Αλλά από τη μία μεριά είναι αυτά και από την άλλη μεριά είναι η πολιτική βούληση να χρησιμοποιείται για στρεβλούς, στρεβλές χρήσεις το σύστημα και σκοπούς. Αλλά υπάρχει και το θέμα της βελτίωσης του συστήματος και της ε, άρσης των ε, αρνητικών συνεπειών για όποιον δεν είναι στο Μητρό. Πρέπει βέβαια να γίνει μια ακριβής σοβαρή αποτίμηση κατάσταση. Είμαι σίγουρο ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Άκουσα του συναδέλφου και εν κατακλείδη πρέπει να σα πω ότι απαιτείται οι ασιατικέ αυτέ χώρε να έχουν την απαραίτητη σχετική πολιτική βούληση. Εμεί δεν μπορούμε να πιέσουμε κανέναν να προβεί σε μεταρρυθμίσει και να χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα, αν δεν θέλει. Τα προγράμματα που σα ανέφερα ήδη έχουν ε, συμφωνηθεί με Ουσμπεκιστάν, με Καζακστάν, με Κυριασία, με Τατζικιστάν. Επομένω υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Πρώτα δεν ξέρω, θέλετε να σας πω και τίποτα άλλο, ό,τι θέλετε στη Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την διαθεσιμότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συζητήσει μαζί μας και να βοηθήσει έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Οι αντιπροσωπείες σε αυτές τις χώρες, ξέρετε, αν είναι ανοιχτές στην κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Θα ήθελα να ζητήσω και από τους συναδέλφους να πάρουν το λόγο. Πρώτα θα δώσω το λόγο στην κυρία Γέγκλε, έμπειρο μέλος της Αντιπροσωπείας για την Κεντρική Ασία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόλις ε, γυρίσαμε από το Καζακστάν και άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που υπόθηκαν σήμερα. Στην αντιπροσωπεία κάναμε μια συνάντηση στο Αλμάτι με τους εκπροσώπους από την ε, χώρα. Νομίζω μία από τους συμμετέχουσες είναι και εδώ σήμερα. Και ε, εκεί χρηματοδοτήσαμε κάποια προγράμματα, το πρόγραμμα Σάν Iraq Μπορέσαμε να δούμε τι γίνεται, μπορέσαμε να μιλήσουμε με τους υπεύθυνου, γιατί το πρόγραμμα αυτό είναι ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο. Ε, και επίσης ε, ε, πήγαμε στην Αστάνα και συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους. Οι εκπρόσωποι της Κομισιόν ήταν εκεί παρόντες και κάναμε πολύ καλές συζητήσεις με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον πρεσβευτή Χιούστον και ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Θα θέλω να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι τα τελευταία χρόνια και, και τα τελευταία δέκα χρόνια πιστεύω ότι όντως προχώρησαν τα πράγματα, υπήρξε πρόοδος και ότι εδώ έχουμε την καλή διάθεση να βοηθήσουμε. Το πρόβλημα τώρα της καταχώρησης ε, είναι σαφές, το γνωρίζουμε. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι η καταχώρηση ε, ε, παντού γίνεται και εμείς θα κάπου. Δεύτερον, πώς γίνεται η καταχώρηση, υπάρχει τρόπος σωστός να γίνει και επίσης το θέμα της διαφθοράς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα όταν χρησιμοποιεί κανεί την καταχώρηση για την πρόθεση της διαφοράς. τότε ναι θα πρέπει να τεθούν ερωτήματα. Στο Αλμάτι και αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με, την, με ευρωπαϊκά χρήματα και μας άφησε πάρα πολλά ερωτήματα. Στην αντιπροσωπεία λοιπόν θα το συζητήσουμε ενδελεχώς και θα ζητήσουμε ερωτήσεις, ε, απαντήσεις και από την Κομισιόν. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος δεν ήταν παρόντες, παρόλο που είχαμε ζητήσει από πριν, από πολύ πριν, να είναι εκεί παρόντες. Δεν τα καταφέραμε. Οι δύο εκπρόσωποι μπόρεσαν, μάλλον δεν μπόρεσαν, να απαντήσουν σε καμία από τις ερωτήσεις μας. Ό,τι μας είπαν ήταν στα ρώσικα. Δεν είχαμε καμία παρουσίαση, καμία πληροφόρηση στα αγγλικά. Μας ζητούσαν συνεχώς το κοινοβούλιο να δεσμευθούμε ότι οι πολίτες που είναι εκεί στο Αλματί που ζουν σε μια παραγκούπολη που εντάξει δεν είναι το χειρότερο αλλά υπάρχουν και χειρότερα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να νομιμοποιηθούν. Εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα τέτοιο, δεν μπορούσαμε εμείς να αναλάβουμε ένα κομμάτι της χώρας, δεν μπορούσαμε να νομιμοποιήσουμε εμείς ένα κομμάτι της χώρας. Εμείς έπρεπε απλώς να θέσουμε ερωτήματα και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα όπως τα είπε τώρα και ο εκπρόσωπος από την Κομισιόν. Και εμείς θα συνεχίσουμε να ρωτούμε στην ε, αποστολή. Ε, τα, τα χρήματά μας όντως επενδύονται σωστά. Δηλαδή εξεπλάγημεν με την κατάσταση αυτή. Πραγματικά όλοι εξεπλάγημεν. Και γι' αυτό δεν θέλω σήμερα να πω κάτι άλλο. Ε, θα το συνεχίσουμε, θα το παρακολουθούμε και μέσω της αντιπροσωπείας αλλά και μέσω της Κομισιόν. Για την στρατηγική που, ε, παρακολουθούμε εμείς θα πρέπει να μελετήσουμε τα πράγματα πολύ ε, προσεκτικά. Εγώ χαίρομαι πολύ που υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν εξαρτάται και διεξάγεται από την όχι από την κυβέρνηση αλλά από μη κυβερνητικές οργάνωσεις. Παρ' όλα αυτά έχουμε και πάρα πολλά ερωτήματα. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γέγκλε για την παρουσίασή σας. Κυρία Βάιντερ. Πράγματι μαζί με τους βοηθούς μας προσπαθήσαμε να δούμε κάπως τα πράγματα πώς πηγαίνουν. μετά από αυτά που είδαμε μείναμε με πάρα πολλές απορίες. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι λίγο πιο προσεκτική όταν επιλέγει τα προγράμματα τα οποία υποστηρίζουν τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και να αξιολογεί τα προγράμματα αυτά περισσότερο πιο προσεκτικά εν πάση περιπτώσει είχαμε επαφές με νοικιό στην περιοχή και είδαμε ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και σε ε, πολιτιστικά θέματα σε σχέση με τη μεταχείριση των παιδιών, ε, σε σχέση με την ελευθερία του τύπου. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα στο Καζακστάν και το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Γέγκλε προκαλεί πολλά προβλήματα και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά χρήματα για να νομιμοποιούνται παράνομες ενέργειες. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα και θα συμφωνήσω με την κυρία Γέγκλε ότι θα πρέπει να ερευνήσουμε το θέμα σε βάθος και να δούμε ε, ποια είναι τα προγράμματα τα οποία στηρίζονται από ευρωπαϊκά ταμεία. Υπάρχουν 12 εκατομμύρια για τον επόμενο χρόνο, αλλά όπως είπα σε τομείς όπως τα παιδιά, η ελευθερία του τύπου, οι γλώσσες, ο πολιτισμός, μένει πάρα πολλά να γίνουν στο Καζακστάν. Το σύστημα τώρα απογραφής. Εγώ πρωτοέρχομαι από τη Λετωνία και να πω στην εκπρόσωπο του Κυργιστάν ότι η χώρα μου δεν είναι χώρα της ε, Συνομοσπονδίας ούτε και η Εσθονία. Είμαστε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να. Και έχουμε ε, πράγματι ε, γνώση του συστήματος Πραπίσκα και ε, ξέρουμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο θέλει να επιβάλλει εκ των άνω έλεγχο. Βέβαια πρέπει να υπάρξει κάποιος έλεγχος σαν παράδειγμα της μετανάστευσης. Ξέρω ότι δημιουργούνται προβλήματα για την πόλη του Αλμάτι. Έρχονται πολλοί παράνομοι μετανάστες και ε, ζητούν να νομιμοποιηθούν και να νομιμοποιηθεί η παρουσία τους. Εν πάση περιπτώσει οι χώρες της Κεντρικής Ασίας χρειάζονται βοήθεια για το πώς θα περάσουν από το σύστημα πραπίσκα σε ένα πολιτισμένο σύστημα απογραφής και εκεί οι χώρες μας όπως η Εστονία, η Λετωνία και η Λιθουανία, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θυμίζω, μπορούν να βοηθήσουν. Η συνάντηση που συναντήθηκε με τις ΜΚΙΟ στην Αλμάτα ήταν ε, ιδιαίτερα χρήσιμη. Ένας από τους εκπροσώπους αυτής της συνάντησης είναι εδώ. θα προετοιμάσουμε την έκθεσή μας, την έκθεση της αντιπροσωπείας και η βασική ανησυχία η οποία μου έχει μείνει από την επίσκεψη αυτή είναι η ελευθερία του τύπου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις συμπληρωματικές πληροφορίες. Δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο και ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ομιλητές μας και ίσως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Νι. Να διευκρινίσω ένα τμήμα της παρουσίασής μου. Όπως είπα στο Καζακστάν, το σύστημα το οποίο λειτουργεί για την απογραφή ε, δεν έχει σχέση με το σοβιετικό σύστημα της Παπίσκα. Και θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει και πρόβλημα διαφθοράς. Το σύστημα όμως ε, της των κοινωνικών παροχών ε, συνδέεται με το θέμα της απογραφής και όταν οι πληθυσμοί μετακινούνται, οι πολίτες μετακινούνται, ε, δεν μπορούν να καταγραφούν στη νέα περιοχή στην οποία εγκαθίστανται και δεν μπορούν να τύχουν κοινωνικής ασφάλισης, σαν παράδειγμα. Τι κάνει. Αυτή είναι η δυσκολία στην περίπτωση του Καζακστάν, είναι όταν υπάρχουν μετακινήσεις του πληθυσμού ή όταν θέλει να επιστρέψει ο πολίτης σαν παράδειγμα στην περιοχή από την οποία προέρχεται που μπορεί να είναι πολύ μακριά. Είναι ίσως οι αποστάσεις τεράστιες, από τη μία πόλη στην άλλη 2.000 χιλιόμετρα. Και αυτό παίρνει και πολύ χρόνο γιατί δεν έχουμε και καλά συστήματα μεταφοράς. για να μπορέσουν ας πούμε να ζητήσουν βοήθεια από το κράτος ε, για οικιστικούς λόγους θα πρέπει να αποδείξει ο συγκεκριμένος πολίτης ότι έχει ένα πιστοποιητικό και ότι είναι εγγεγραμμένο στη συγκεκριμένη πόλη. Το σύστημα λοιπόν των κοινωνικών παροχών προαπαιτεί θα έλεγα να αποδείξει ο πολίτης ότι είναι εγγεγραμμένο στην περιοχή. Και καλό θα ήταν να γίνει το σύστημα αυτό πιο φιλελεύθερο και θα πρέπει οι αρχές να δέχονται την αίτηση ανεξάρτητα από τον τόπο παραμονής ε, του πληθυσμού. Ζούμε σε ένα σύγχρονο κόσμο και το Καζακστάν μπορούν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Το θέμα είναι ότι οι δημόσιες αρχές εμένουν στα γραφειοκρατικά απαιτούμενα και δεν βοηθούν έτσι εκατοντάδες χιλιάδες ε, κάτοικοι του Καζακστάν είναι εκτός συστήματος κοινωνικής προστασίας για τέτοιους τυπικούς λόγους. Πρέπει λοιπόν να εντοπίσουμε τα πρόσωπα αυτά, να δούμε ακριβώς ποιοι χρειάζονται κοινωνική προστασία και να τους την δώσουμε. Ευχαριστούμε για όσα μας εξηγήσατε, λέει ο Πρόεδρος. Αλλά και η κυρία Γιακουμπόβα, φαντάζομαι θέλει το λόγο, η κυρία Νιαζόβα. Yeah, um, ναι, Πρόεδρε. Αυτό θα σα πω ότι έχουμε εδώ μαζικέ πράγματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουσβεκιστάν. Και αυτό όχι διότι δεν υπάρχουν τα χρήματα ή οι δυνατότητε γενικότερα, αλλά διότι απουσιάζει η πολιτική βούληση. Δεν χρειάζεται να δώσετε χρήματα στο, στην κυβέρνηση ή να εκπαιδεύσετε κανέναν για να σταματήσουν τα, βασανιστήρια. Δεν υπάρχει ελευθερία λόγου, διότι δεν υπάρχει. Δεν θα υπάρχει πολιτική βούληση. Γι' αυτό σας λέω. Όταν πιάσει τόπο το πρόγραμμα για το κράτος δικαίου, τότε θα δούμε αποτελέσματα. Μα τι, τι, τι, να, τι, τους δημοσιογράφους οι οποίοι Κατά εκατοντάδες φυλακίζονται. Χαμένα χρήματα θα είναι. Για το αρχείο αυτό την υποχρέωση εγγραφή στο Μητρό τα πράγματα διαφέρουν από μια χώρα στην άλλη. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορεί κανείς χωρίς κρατική άδεια να ταξιδέψει από τη μια χώρα στην άλλη. Ακόμα και αν έχει τα προσόντα, προσληφθεί κάπου, ακόμα και αν έχει που να μείνει θα πρέπει να πάρει επίσημη άδεια για να μετακινηθεί από το ένα χωριό στο άλλο και δεν μιλάμε για λοδαπούς, μιλάμε για τους Ουσμπέκους, οι οποίοι μέσα στο Ουσμπεκιστάν ε, έχουν περιορισμό μετακίνησης. Την ίδια του τη χώρα. Ευχαριστούμε κύριε Νιαζόβα. Λέει πρόεδρος. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να λάβει το λόγο για τα όσα ακούστηκαν τώρα για το Καζακστάν ειδικότερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες του να υλοποιήσουμε πολλά από αυτά τα προγράμματα που έχουμε εξαγγείλει δεν θέλουμε ακριβώς να έχουμε όλα αυτά τα σεμινάρια για κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι τελικά πρόκειται να φυλακιστούν. Οπότε τώρα αυτό λέμε στις κυβερνήσεις της περιοχής ότι θα πρέπει να στάσουν προσοχή τους στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Βεβαίως και κάποια από αυτά τα προγράμματα τελικά δεν πρόκειται να αρχίσουν να τρέχουν ποτέ. Γιατί δεν θα πληρούνται τα σχετικά κριτήρια. Αυτό είναι γνωστό. Θα, πρέπει να τρέξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πιάσει τόπο για να μην πάνε χαμένα τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Φυσικά και δεν ε, αποδίδουν το ίδιο όλα τα προγράμματα, δεν λειτουργούν το ίδιο καλά και προσπαθούμε να το φροντίσουμε. και όπως ε, είπε κάποιος βουλευτής με τίποτα δεν θέλουμε με τα κοινωτικά χρήματα να νομιμοποιήσουμε κάποιες ε, καταστάσεις που αποτελούν εγκλήματα. Άρα, θα έρθουμε σε επαφή με τις ε, γιατί με την αρμόδια κυβέρνηση, διότι πάντοτε Όπω γίνεται παντού στον κόσμο υπάρχει αυτού του είδους η εμπλοκή μη κυβερνών οργανώσεων, να ακουστούν όλες οι απόψεις. Αυτό και είπα στους ε, εκδεξιών μου Συναδέλφου που θα πρέπει να σε επαφή με τις ε, αντιπροσωπείες που είναι και οι αρμόδιοι για τη διάρθρωση του προγράμματος. Όπως είπαμε προηγουμένως, θα πρέπει να εξετάζεται η κατάσταση ε, και να λαμβάνεται υπόψη πραγματική διάσταση των γεγονότων, γιατί μόλις πριν από μία τριετία δεν μπορούσαμε καν να θέσουμε αυτά τα θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων ε, στις συναντήσεις με τους ε, υπουργούς εξωτερικών αυτών των χωρών. Τώρα όμως θα συζητάμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το έχω ακούσει εγώ με τα αυτιά μου γιατί έχω παραστεί σε τέτοιε επαφέ. Γιατί ο Τάδε βρίσκεται στη φυλακή. Πολύ συγκεκριμένα. Όσο βέβαια είναι δύσκολη η συνεννόηση. Αλλά έχουμε αποσπάσει αποτελέσματα. Βεβαίω. Πάντοτε υπάρχει αμοιβιότητα. Και φυσικά και είμαι αισιόδοξο, αν δεν είμαι αισιόδοξο θα είχα παραιτηθεί. Αλλά όσο και να είναι δύσκολη αυτή η προσπάθεια προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα στους Ασιάτες ότι δεν τους υποτιμούμε. Από την άλλη μεριά, αντίθετα, είναι σεβαστές οι ευρωπαϊκές αξίες. Ακούγεται η φωνή μας. Όταν τους μιλούμε, μας ακούν. Ελπίζουμε πάνω όλα καλά. Ευχαριστούμε εμείς, λέει η Πρόεδρος, και εδώ στο λόγο στην κυρία Γέγκλε, και κατόπιν θα έχουμε την Απρολέθ και κάποιον προσπαθεί να λάβει το λόγο. Γέγκλε. Με αυτή την ε, ευκαιρία θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πλησιώσουμε όπως γίνει καλύτερη την προσωπία μας και στο ε, Καζακστάν αλλά και στο Ουσβεκιστάν. ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια με κάποιες δυσκολίες. Όμως, στη συνέχεια, η δουλειά μας έπιασε τόπο. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει τα πράγματα. Έχετε το λόγο στα ρωσικά. Μπορώ να μιλήσω ρωσικά, δεν είναι, ναι. Για το Κυριεστάν θέλω να σας πω. Θα ήθελα να μου πείτε σε σχέση με την Υπουργική Σύνοδο πότε προβλέπετε να γίνει ακριβώς. Επίσης, τι γίνεται με αυτή την πρωτοβουλία όσον αφορά τη θέσπιση κάποιων ειδικών μέτρων, όσον αφορά την προπίσκα, δηλαδή αυτό το σύστημα της ε, δήλωσης στο Μητρό. Τι θα γίνει στην Υπουργή Συνόδο, θα συζητηθεί. Επιτροπή. Ναι, για την Υπουργική Συνάντηση. Έχω να σας πω ότι συστηματικά σε κάθε Υπουργική Σύνοδο συζητείται η πολιτική κατάσταση σε διμερές επίπεδο και στο σύνολο της περιοχής. Συστηματικά και με τις πέντε χώρες που κάνουμε αυτό. Τουρκμανιστάν, Ουσμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Χιργισία, Καζακστάν, όλες, όλες. Και συμφωνούμε τι θα συζητηθεί στη Μεσή Διαταξή. Ανεξαρτήσεις δικαιοσύνη, φυλάκιση δημοσιογράφων, καταστολή ε, εις βάρος των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά συζητούνται. Και όπως προείπα, συζητούνται και ατομικές περιπτώσεις. Βέβαια, όταν γίνεται μια συνάντηση σε μια ώρα ή μια μισή ώρα, πρέπει να καλυφθούν πολλά θέματα. Πολλά θέματα και όχι μόνο η πολιτική κατάσταση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορούμε να συζητήσουμε, ας πούμε, για θέματα περιβάλλοντος, ε, θέμα ε, υδάτων Αλλά πάντως αυτά τα θέματα που είπατε τα συζητούμε συστηματικά. Τώρα, για το σύστημα της προπίσκα και τις συνέπειές του, επίσης, το θέμα αυτό έχει ζητήσει σε όλες αυτές τις χώρες στα πλαίσια του διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι ω επιτοπλίστων αυτό ιδίω σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Γιατί όταν λέμε για κάποιον ο οποίο ε, θα πρέπει ελεύθερα να μετακινηθεί από μια χώρα, από μια πόλη στην άλλη στην ίδια χώρα, θα πρέπει να ζητηθεί και στι λεπτομέρειε το οποίο απαιτεί χρόνο. Αλλά χρειάζεται και ειδικού. Βυρογνώμονε. Δεν είναι δυνατόν ε, ένα υπουργό ε, από τη μία και από την άλλη μεριά να κάθεται και συζητούν τι λεπτομέρειε αλλά στην Υπουργική Σύνοδο συζητείται το θέμα επί της αρχής και ε, για τις λεπτομέρειες συζητείται αυτό στο διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πότε και έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και τις ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και την Απερντεύ και τη Κομισιόν που για αυτή την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων η οποία ελπίζω να οδηγήσει και σε καλύτερο συντονισμό και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αντιστοίχως στις δικές σας χώρες. Για μας, την Υποεπιτροπή, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε για το πώ οι αντιπροσωπείε συμπεριλαμβάνουν την κοινωνία των πολιτών στην καθημερινή του δουλειά και πώ ενημερώνουν την κοινωνία των πολιτών για το τι γίνεται με τι κυβερνήσει και με τι δραστηριότητε του. Όλοι λοιπόν πρέπει να έχουμε μια στρατηγική συγκεκριμένη για τα θέματα τη κοινωνία των πολιτών και, της, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στην Ουάσιγκτον και η αντιπροσωπεία έχει ένα σημείο επαφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, έναν υπάλληλο. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει σε όλες τις αντιπροσωπείες. Οπότε θα συνεχίσουμε να το συζητούμε για να δούμε πώς μπορεί το Κοινοβούλιο να βοηθήσει. Είναι πολύ ενθαρρυντικό όμως που η Κομισιόν έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ και την κυρία Γκέγκλη και την κυρία Βαϊντέρα. Ο κύριος Σούστερ τώρα από την Άπροντεβ. Α, εκεί στο βάθος είστε, μάλιστα. Κυρία Χάουταλα, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να μας, που μας δίνετε την ευκαιρία να θέσουμε αυτό το θέμα μαζί με τους αδέλφους μας για τα δικαιώματα στην Κεντρική Ασία. Έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πολιτική βούληση στις χώρες αυτές της Κεντρικής Ασίας για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Για την, ε, τώρα για την αντιπροσωπεία που πήγε στο Καζακστάν αναρωτιέμαι αν χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να ενθαρρύνει την ύπαρξη πολιτικής βούλησης Ακούω εδώ τους εκπροσώπους της κυβέρνησης του Καζακστάν όταν ας πούμε συμφωνείς τόσο γρήγορα για το ότι οι άνθρωποι ε, εκμεταλλεύονται τη γη που δεν είναι δική τους αλλά δεν ρωτάς γιατί την εκμεταλλεύονται και γιατί δεν μπορούν να την αγοράσουν αυτή τη γη που θα ήθελαν ίσως γιατί δεν είναι καταχωρημένοι, αν δεν θέσεις αυτά τα ερωτήματα, τότε δε, πώς θα δημιουργήσεις και πολιτική βούληση. Ευχαριστώ. Mrs. says that this has been done. So, uh, thank you for APRODEV and uh, thank you for everyone. Ευχαριστώ. για την συμμετοχή σας. Η Κεντρική Ασία πάντα είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας. Πάντα. Uh, το 7 δεν το έχουμε να το συζητήσουμε γιατί ο κύριος Μάρτιν δεν μπορεί να ήταν μαζί μας σήμερα. Και το σημείο 8, για το σημείο 8 τώρα, θα πρέπει να διακόψουμε λίγο έτσι ώστε να μπορέσουν να φύγουν αυτοί που είναι εδώ για τα της Κεντρικής Ασίας πριν περάσουμε στο θέμα για τους ηθαγενείς πληθυσμούς.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 Μπορούμε τώρα να ακούσουμε από την αντιπροσωπεία για, τα, για το φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα του, του ΟΗΕ για τους αυτόχθονες από τις 28 στις 30 Απριλίου στην Νέα Υόρκη έγινε το φόρουμ και χαίρομαι που είναι διάφορα μέλη της αντιπροσωπείας εδώ και μέλη της Επιτροπής μας βεβαίως. Um, πολύ χρήσιμη ήταν αυτή η αποστολή της αντιπροσωπείας, οπότε τώρα θα δούμε ποια είναι και τα αποτελέσματα και τι έχουν να πούνε τα μέλη της αντιπροσωπείας. Είναι εδώ ο κύριος Πρόντι, η κυρία Κιλ Νίλσεν και η κυρία Γιάστραμ. Και ο κύριος Πόγκα επίσης είναι εδώ. Οπότε πώς να σας δώσω το λόγο, με ποια σειρά θέλετε. Ο κύριος Πρόντι να ξεκινήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την δυνατότητα που μου δίνετε. Νομίζω ότι ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα στα πλαίσια της συμμετοχής της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο μόνιμο ε, φόρουμ για τα προβλήματα των Ιθαγενών ε, λαών. Το ενδιαφέρον μου αφορά κυρίως την πλαισίωση θα έλεγα του προβλήματος της υπερθέρμανσης και της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκαλεί η υπερθέρμανση και ότι έχει σχέση με την πολιτική, θα έλεγα, που εμπλέκει άμεσα τους ηθαγενείς ε, πληθυσμούς και το θέμα της ρέντα. Τη μείωση δηλαδή των εκπομπών ε, αερίων θερμοκηπίου από την υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος. Ε, percezione è stato molto importante anche eh, in particolare per quanto riguarda eh, eh, δώσαμε ειδική προσοχή στον τρόπο που ανταλαμβάνονται ή αντιλαμβάνονται συγγνώμη, οι ηθαγενείς πληθυσμοί το πρόβλημα και το θέμα της ανταλλαγής των ποσοστώσεων. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στην δήλωση της Κοτσαμπάμπα ήταν αυτός ο φόβος ο οποίος υπάρχει για να γίνει για την ατμόσφαιρα αυτό το οποίο έχει γίνει για τους υδάτινους πόρους, δηλαδή μία μορφή ιδιωτικοποίησης του αέρα. Η αντίληψη αυτή είναι θα έλεγα σαφής σε ορισμένες από τις πληθυσμιακές αυτές ομάδες και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αρχίσει να μας ανησυχεί. Εγώ πήρα μέρος στην Ολομέλεια, στη συζήτηση της Ολομέλειας και ζήτησα να διαβεβαιώσω τους πληθυσμούς αυτούς ότι αυτή η αγορά, όπως θα έλεγε κανείς, των εκπομπών των εκπομπών ε, αυτών δεν είναι ένα βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της ατμόσφαιρας που αναπνέουμε αλλά είναι ένας τρόπος μέσα από τον οποίο προσπαθούμε να αξιολογήσουμε την αποζημίωση την οποία θα πρέπει να δώσουμε στις χώρες οι οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν τις, ε, τα, τις δραστικές τους εκτάσεις κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η, το εμπόριο αν θέλετε αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει έμεσα και σαν πολιτιστικός φύλακας στον κόσμο σήμερα και σαν μια δυνατότητα εγγύησης θα έλεγα της κληρονομιάς της ανθρωπότητας και όλες αυτές οι υπηρεσίες τις οποίες μπορεί να προσφέρει ε, ε, το, το κλίμα ε, και οι αλλαγές σε μια σφαιρική πολιτική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται και σαν μια αναγνώριση θα έλεγα της ίδιας της αξίας αυτών των ηθαγενών λαών και να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τους ηθαγενείς λαούς έτσι ώστε να διατηρήσουμε και όχι μόνο το περιβάλλον τους αλλά τον πολιτισμό τους και φυσικά τον χώρο μέσα στον οποίο ε, ζουν. Νομίζω ότι η παρουσία μας εκεί ήταν ιδιαίτερα εμπλουτιστική Ενθυμούμε μια μεγάλη συζήτηση την οποία είχαμε με τον πρέσβη Παύλο Σορών της Δημοκρατίας ε, της ε, Βολιβίας εκμεταλλευόμενος και την δυνατότητα που είχαμε σε μη επίσημο επίπεδο να έχουμε επαφές οι οποίες ήταν νομίζω και αυτές πολύ απαραίτητες επαφές που μας επέτρεψαν να κατανοήσουμε περισσότερο τα αιτήματα των ηθαγενών και να εμπλέξουμε τους πληθυσμούς αυτούς στην αναζήτηση των προσπαθειών ε, επίλυσης των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε παγκόσμια πλέον. Ευχαριστώ κύριε Πρόντι για μια ενδιαφέρουσα ε, συζήτηση. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Κιλ Νίλσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι το θέμα της προέσπισης των δασών της ε, εμπορίας ε, των ε, αερίων θερμοκηπίου και τα λοιπά και του συστήματος εμπορίας αυτού θα ήθελα να πω ότι είναι κάτι το οποίο δημιουργεί κάποια σύγχυση σε ορισμένους πληθυσμούς ιδιαίτερα αυτοί που προέρχονται Αμερική. Εκφράζουν τη λύπη τους που δεν ακούστηκε η άποψή τους για την επεξεργασία αυτής της διαδικασίας και θεωρούν ότι τίποτα δεν δίδει εγγυήσεις ε, για τα συμφέροντά τους και καταγγέλουν εν πάση περιπτώσει το θέμα της εμπορικής αντιμετώπισης του προβλήματος μέσω της ε, πλήρους ε, εμπορικής αντιμετώπισης των δασών. Για αυτούς το δάσος έχει μια διανοητική πνευματική διάσταση και θέλουν να μην αντιμετωπίζουμε το δάσος σαν κάτι το αυστηρά οικονομικό. Το δάσος για αυτούς είναι μια θα έλεγα αξία πνευματική και όχι εμπορική. Έχουν αμφιβολίες λοιπόν για το σύστημα της αγοράς το οποίο επιτρέπει να εξαγοράζουμε τις δικές μας συνειδήσεις αλλά δεν μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων και δεν διαβεβαιεί σε καμία περίπτωση ε, τους ηθαγενείς των αγώνα που δίνουν για επιβίωση. Ο Τζον Κάρλινγκ, ο οποίος εκπροσωπεί τις Φιλιππίνες, είχε μια αντίληψη κάπως πιο μετριοπαθή γύρω από το θέμα το συγκεκριμένο και πιστεύει ότι σε σχέση με το RED θα πρέπει να δούμε ε, ε, πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε και δεν το αμφισβητούσε πλήρως για τις αυτόχθονες κοινότητες των Φιλιππινών όταν ε, είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στην απώλεια των δασών υπέρ του εμπορίου μέσω της εκμετάλλευσης ε, των φραγμάτων κτλ ή της διατήρησης μέσω του μηχανισμού του ΡΕΝΤ προφανώς προτιμούσε το ΡΕΝΤ. Γι' αυτό λοιπόν η συζήτηση ήταν σαφής. Εγώ ξέφρασα την απογοήτευσή μου για την υπερεκπροσώπηση των πληθυσμών της Λατινικής Αμερικής κάτι το οποίο έχει σχέση περισσότερο με την παρουσία, την, τέλεση, την οργάνωση του συγκεκριμένου φόρουμ στις Ηνωμένε Πολιτείες. Δεν συναντηθήκαμε σαν παράδειγμα με εκπροσώπους λαών, φυλών που ζουν στην Αφρική Ίσως θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στο πού θα μπορούσε να συνεδριάζει ένα τέτοιο φόρουμ, ένα φόρουμ που θα συνεδριάζει στη Γενέβη, σαν παράδειγμα, ίσως να επιτρέψει να εκπροσωπηθούν αντιπροσωπευτικότερα. Ο κύριος Αχμέντ Μοχάμεντ που εκπροσωπεί του Σαματσίγκ του Νότου του Μαρόκου πήρε το λόγο και αναφέρθηκε ε, στις διεκδικήσεις ε, των πληθυσμών αυτών που φύγονται άμεσα από την ε, υπερθέρμανση και την απερίμωση. Υπήρξε επίσης μια σημαντική εκπροσώπηση του Φόρουμ του Νεγκεύ για την ισότητα των πολιτών καταγγέλθηκαν ε, τα, ε, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Βεδουίνων στην έρημο του Νεγκέβ στο Ισραήλ. Όπως επίσης ε, και της Μονίκ από την Ταϊτή που εκπροσωπεί συλλόγους που καταπολεμούν τις αρνητικές επιπτώσεις του ελέγχου του γαλλικού κράτους ζητώντας ε, η ε, γαλλική πολυνησία να επανέλθει στον κατάλογο των χωρών που θα πρέπει να αποαπικιοποιηθούν. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ε, πολύ ενδιαφέρον και εγώ προσωπικά σε, μια συγκεκριμένη, σε ένα συγκεκριμένο γαλλικό νομό στην Γουιάννα, Γουιάννα γαλλική, ε, εγώ εξέφρασα τη λύπη μου για την πλήρη απουσία των εκπροσώπων αυτών των Ινδιάνων της Γουιάνας. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι αυτοί πολίτες να συμμετέχουν στα φόρα αυτά στο μέλλον. Ξέρω ότι για οικονομικούς λόγους δεν μπόρεσαν να κάνουν τη μετακίνηση αυτή και λυπάμαι γι' αυτό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα λοιπόν που αφορούν τους ευρωπαϊκούς αυτόχθονες ε, ε, ε, πληθυσμούς. Υπήρχε βέβαια εκπρόσωπος ε, των Ινουίτ, αλλά δεν υπήρχε εκπρόσωπος των Γάλλων Ινδιάνων της Γαλλικής Γουιάνας που είναι θύματα μιας παράνομης εκμετάλλευσης των, του χρυσού στη χώρα αυτή και ε, αυτοί αναγκάζονται αντί να ψαρεύουν ψάρια πλέον και να καταναλώνουν ψάρια όπως πάντα το έκαναν από τα ποτάμια τους αναγκάζονται να τα καταναλώνουν με πολλά δηλητήρια γιατί υπάρχει η παράνομη ε, ε, χρυσορυχία η οποία προηγείται. Τίποτα περισσότερο. Κύριε Αγγελίνη, σας ευχαριστώ με μεγάλη μας χαρά. Ακούσαμε να αναφέρετε τους Ευρωπαίους ηθαγενείς γιατί ασχολούμαι με τους Σάμι πολλά χρόνια. Όπως ξέρετε, δεν έχει προσχωρήσει στις συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας η Φιλανδία σε σχέση με την κτήση γης από αυτούς και έχουμε συνεχείς προστριβές μεταξύ αυτών, των Σάμι και της κυβέρνησης που είναι ο κύριος αυτών των γεών. Άλλοι Δύο συνάδελφοι μέλη στην προσωπία στέλνουν το γνώμη και μεγάλη μου χαρά το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Μιλήσατε και για τους Ευρωπαίους ή Ιθαγενείς. Όλοι ήμασταν ε, εκεί. Ε, είναι θέμα που δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ο συνάδελφος ήδη είπε ότι πρέπει να είναι στο κέντρο των προσπαθειών μας ναι, οι ηθαγενείς της ε, Νοτιοαμερικής. Πρέπει όμως να δούμε και λίγο πέρα από αυτό. Νομίζω ότι μάλλον ήταν η πρώτη φορά που ήμουν σε μια τέτοια διάσκεψη και θα πρέπει μάλλον να θέσουμε και το ερώτημα Καταρχήν, εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα να, που το ζήσαμε όλο αυτό, αλλά θα πρέπει να θέσουμε ένα ερώτημα που ίσως να είναι και τυπικά ευρωπαϊκό. Ε, και πού θα καταλήξει όλο αυτό. Δηλαδή, όλο οι σωστοί άνθρωποι είναι σε τέτοιες διασκέψεις και παρακολουθούν και εξάγουν συμπεράσματα. Εντάξει, είναι καλά όλα αυτά. Είναι καλό οι λαοί που πλήττονται να μπορούν να μιλήσουν και να μας πούν ποια είναι τα προβλήματά τους, αλλά το πιο σημαντικό είναι η υπεύθυνη πολιτική, ο καθένας στον τομέα του, να προσπαθήσει να δράσει. Και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω να συνεχίσουμε να στέλνουμε αποστολές και ad hoc αντιπροσωπείες σε τέτοιες ε, ε, διασκέψεις και να παραμείνουμε στο διάλογο, να δούμε σε ποιους τομείς υπάρχει δυνατότητα για κάποιο χειρισμό, πού μπορούμε να στηρίξουμε εμείς την όλη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Δηλαδή στο τέλος Αξιέμεινε έτσι ένα άσχημο συνέστημα γιατί ωραία, τα είπαμε όλοι πολύ ωραία αλλά τελικά δεν γίνονται και πολλά και νομίζω ότι ε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους ε, προστατεύσουμε γιατί πραγματικά η αδικία πλήττει αυτές ακριβώς τις κοινότητες. Ευχαριστώ. Thank you, Κυρία Σνίμπερ, σας ευχαριστώ. Όταν χειρώ των συμπερασμάτων θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε και αυτό το οποίο είπατε. Εκτός βέβαια κάποιος θέλει να απαντήσει. Κύριε Μπόγκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά συμμετέσχουν στην αντιπροσωπεία. Και όταν συναντήσαμε τον ε, πρέσβη στη Νέα Υόρκη το είπα ότι είμαι και εγώ ηθαγενής, αυτόχθον, που όμως κατοικώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είμαι απέναντι όσον αφορά τους αυτόχθενες που, και τις διεκδικήσεις τους. Κάποιες διευκρινήσεις δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε τέτοιες συναντήσεις γιατί έχω συμμετάσχει στην ε, Επιτροπή για την αυτοδιαχείριση και πάυση της απεικιοκρατίας. Τα πιο σημαντικά τα οποία προτάσουν σε επιχειρήματα αυτοί αυτόχθονες είναι το τι θα γίνει με τα δάση τους. Δηλαδή μιλούν για τις συνέπειες αλλαγής του κλίματος. Διότι εκεί που κατοικούν δεν προπονούνται πολύ, αλλά όπως είπε ο κύριος Πρόντι, αυτοί μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι οι, οι φύλακες αυτού του παγκόσμιου πολιτισμού. Υπάρχουν όμως κάποιες, ε, ε άλλες, ε, κάποια άλλα θέματα όπως η οικονομική ανάπτυξη αλλά οι βασικές διεκδικήσεις αυτών των ανθρώπων είναι το τι θα γίνει με το μέρος που ζουν. Και εμείς που είμαστε μεγάλα κράτη ευρωπαϊκά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ε, αυτοί οι περιορισμένοι στον αριθμό τι θέλουν. Συμφωνώ βεβαίω με αυτές τις διεκδικήσεις, είναι πολιτικές διεκδικήσεις τους για το καθώς θα τους διέπει σε σχέση με την κυβέρνηση του κράτους όπου κατοικούν κλπ. Οπότε θα πρέπει κανείς με σοφροσύνη να, να δει πώς ε, θα χειριστεί αυτές τις διεκδικήσεις αλλά θα πρέπει να εξεταστεί επίσης τι γίνεται με τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις των σχετικών διασκέψεων και συνδιασκέψεων. Γιατί γίνεται κάποια πρόοδος, αλλά δεν είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά τα ψηφίσματα, τις αποφάσεις των σχετικών οργανισμών και το αυτών των συναντήσεων. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κύριε Μπόγκα, ευχαριστούμε εμείς. Θα ήθελε κάποιος να κάνει μια σύνθεση όσον αφορά αυτά τα οποία αναφέρθηκαν. Κύριε Κιλνίλτσα. Όχι, απλώς θα ήθελα συμπληρωματικά να σας ε, αναφέρω ε, πάνω στο θέμα των δασών είναι ότι το φόρουμ που θα γίνει του χρόνου θα ασχοληθεί ειδικά με αυτά τα δάση. Άρα αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα στο φόρουμ του χρόνου. Κάποιο άλλο ή θέλει το λόγο. Και εγώ λέει πρώτα θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο είπε θα ήθελε το λόγο. Α, και εγώ λέει πρώτος θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο είπε η κυρία Κυρνίλσεν για αυτούς τους ε, πληθυσμούς της Δυτικής Παππού. Έγινε μια συζήτηση της μάκρον όσον αφορά την απερίμωση των δασών, την καταστροφή των δασών, ε, αυτές τις ε, φοιτίες, τα το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων και ακούσατε για τη συνεργασία Ινδονησίας-Νορβηγίας. Οπότε είχαμε και αυτό το πάγωμα, το μορατόριο της καταστόλης των δασών για κάποια χρόνια και το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί τέτοιες πρακτικές καταστρέφουν όπως ο κύριος Πρόντι και το κλίμα αλλά απειλούν και αυτούς τους πάρα πολύ σημαντικούς πληθυσμούς. Παντού. Τώρα καταλαβαίνουμε καλύτερα τότε θα πρέπει να ξεχνούμε εδώ στο έργο μας για ανθρώπινα δικαιώματα τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Να το έχουμε στο μυαλό μας συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο ίσως δεν το έχουν προσέξει τόσο πολύ και ελπίζω ότι θα επανέλθουμε όσον αφορά το τι θα γίνει και αν κάνω λάθος διορθώστε με στην Ευρώπη έχουμε τους Σάμι μόνο τους Σάμι έχουμε σαν αυτόχθανα τέτοιο πληθυσμό Α, είναι υπεράκτια, υπεράκτια επικράτεια. Όχι, δεν, δεν ισχύει αυτό. Τέλος, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για το εξαιρετικό κείμενο αυτό θα πρέπει να παρακολουθήσουμε να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις προτάσεις της αντιπροσωπείας σας και Εδώ μπορούμε να κληρώσουμε την συνεδρίασή μας αφού δεν πρόκειται να γίνει συζήτηση του κ. Μάρτιν. Η δε επόμενη συνεδρίαση είναι την επόμενη εβδομάδα, την 5η στις 9 το πρωί. Θα έχουμε συζήτηση με την Ισπανική Προεδρία. Για να ακούσουμε το δικό συμπεράσμα όσον αφορά τι προσπάθειε που έδωσαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οπότε μην το ξεχνάτε. Και θέλω να σα αναφέρω ότι ο πρόεδρος Μπούζεκ συμφώνησε να έρθει να μας μιλήσει. Όπως ξέρετε είναι πολύ δραστήριος, ενδιαφέρει την ανθρώπινη δικαιώματα ο πρόεδρός μας, οπότε υπάρχει λόγο να ε, τα λέμε και είναι μια ημερομηνία που δημιουργεί κάπως ένα πρόβλημα ε, να σας τα πω και, για να, και να το σκεφτείτε αν μπορείτε να έρθετε 3 ώρες 24 Ιουνίου το πρωί της ίδιας μέρας θα έχουμε συνεδρίαση της υποεπιτροπή μας αλλά σας το λέω για να μου πείτε πόσοι από εσά μπορείτε καλά θα το δούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο άμεσο μέλλον. Γιατί είναι μια ευκαιρία που πρέπει να τη χάσουμε. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη.